συμπεράσματα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 23 Σεπτεμβρίου 2015, δηλώσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη Επιτροπή. Κανονικά θα έπρεπε να δώσω το λόγο τώρα στον πρόεδρο του Συμβουλίου, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι καθοδόν ακόμη. Θέλετε να ξεκινήσετε εσεί, κύριε Γιουνκέρ. Να μην ε, ξεσπάσει όμω καμιά μεγάλη διπλωματική κρίση, έτσι. Για να δούμε άλλη μια φορά πώ έρχεται. Από ό,τι καταλαβαίνω, σε μερικά δευτερόλεπτα θα είναι εδώ. Herr Juncker, stimmt es eigentlich, dass Sie heute Morgen hier auf diesem Platz gesessen haben? Εσείς έχετε έρθει για πόσες φορές εδώ πέρα. Κοιτάξτε, πέντε φορές έχω εκλογεί ευρωβουλευτής, λέει ο κύριος Γιουνκέρ, αλλά η μοίρα με έστειλε με άλλα καθήκοντα εδώ. Ich traue mir das auch zu και πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Ναι, και εγώ μπορεί, θα μπορούσα να είμαι στη θέση σας, κύριε Γιουνκέρ, λέει ο πρόεδρος. Καλά, ας μην αρχίσουμε αυτές τις ε, παρομοιώσεις. Καλώ, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, ξεκινούμε τη συζήτηση για τα συμπεράσματα του Άτυπου Συμβουλίου της 23η Σεπτεμβρίου 2015. Μέχρι να έρθει ο κύριο Τούσκ στον κύριο Γιουνκέρ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καλό είναι να ξεκινάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτη να ομιλεί πριν από το Συμβούλιο, πριν από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Και αυτό θα ήθελα να το ελπίσω και να το διεκδικήσω, αλλά τέλο πάντων αλλιώ θα ήθελε η μοίρα. Κύριε Πρόεδρε. Είχαμε τη συζήτηση 23 Σεπτεμβρίου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους ε, πρόσφυγες και τη μετανάστευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα το θυμάστε ασφαλώς και από το Μάιο, θα έχει μείνει ζωντανό στη μνήμη σας, είχε καταθέσει προτάσεις στο Συμβούλιο, το οποίο χρειάστηκε πολύ περισσότερο χρόνο για να καταλήξει συμφωνία για τις ε, προτάσεις αυτές. Εμείς θα προτιμούσαμε ως Επιτροπή να είχε ομόφωνα λάβει την απόφαση για την αλληλέγγυα κατανομή του αριθμού των προσφύγων στα κράτη-μέλη το Συμβούλιο. Αυτό και για λόγους περισσότερο εσωτερικής πολιτικής και δεσμεύσεως εσωτερικής πολιτικής δεν κατέστη δυνατόν. Και δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου σε τελευταία ανάλυση. Η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο τρόπος με τον οποίο ε, διατυπώθηκε και ε, ορίζει ως κύρια μέθοδο την κοινοτική μέθοδο για τα θέματα αυτά και έτσι αποφάσισαν και οι Υπουργοί με την κοινοτική μέθοδο. Διοργανικά και ως προς τον τρόπο εργασίας, το ότι ελήφθηκαν με αυτόν τον τρόπο η απόφαση είναι καλό σημάδι. Donald Θέλεις να λάβεις το λόγο ή να συνεχίσω. Μια και ήρθες. Βλέπω με, με χαρά ότι έδειξε μεγάλη ευαισθησία το Συμβούλιο. Έγινε η ε, περαιτέρω συζήτηση τώρα και τελικά η απόφαση ελήφθη με την κοινοτική μέθοδο. Τώρα καλό θα ήταν να μην πέσουμε στο βάλτο των αλληλοκαταγγελιών και αλληλοκατηγοριών. Θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα υλοποιηθούν οι αποφάσεις πάνω απ' όλα και αυτό το πράττουμε με, το ταχύτερο, με τη μεγαλύτερη ταχύτητα στα γαλλικά. Εμείς ως Επιτροπή δράσαμε με τρόπο γαλήνιο και κανείς δεν το περίμενε. Είχαμε στις 23 Σεπτεμβρίου το Συμβούλιο, προτείναμε στα θεσμικά όργανα, στις, στα δύο σκέλη δηλαδή α, ε, της δημοσιονομικής διαδικασίας της ε, προτάσεις μας, τις σχετικές με το 2015 και για το 2016 που θα καταθέσουμε εις επόμενες εβδομάδες ε, καταθέσαμε τις προτάσεις για 800 εκατομμύρια. Καταρχάς και με χαρά διαπιστώνω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πάλι κατέστησε δυνατόν ότι θα λάβει απόφαση ταχύτατα. Στις 8 νομίζω του μηνός σε επίπεδο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και στις 15 στην Ολομέλεια. Δηλαδή το Κοινοβούλιο ε, ενστερνίζεται αυτά τα καθήκοντα και την εντολή που έχουμε και εμείς αναλάβει και συμμετέχει ε, στη διαδικασία για την αλληλέγγυα κατανομή του αριθμού των προσφύγων στις χώρες. Πράγμα το οποίο υποχρεώνει και το Συμβούλιο να το ακολουθήσει. Ε, φανταστείτε δηλαδή το Συμβούλιο να ακύρωνε με την στάση του την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό και θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε εσά αλλά και σε όλο το σώμα, κύριε Πρόεδρε, για τον τρόπο και πάνω απ' όλα την ταχύτητα με την οποία ε, διαχειριστήκατε το θέμα. Όπω άλλωστε πράττει συχνά το Κοινοβούλιο, πιστεύω ότι θα συμβεί το ίδιο και με τα δημοσιονομικά, γιατί θα πρέπει να ενισχυθούν τα κονδύλια για τη Frontex και την Europol, όπως και για το Ευρωπαϊκό Γραφείο Στήριξης για το Άσυλο. η Επιτροπή έχει να διαθέσει έως και 600 υπαλλήλους για να στηρίξει την Ελλάδα στην προστασία των εξωτερικών της συνόρων με στο άμεσα προσεχές διάστημα. Άρα θα αναπτύξουμε μεγάλο δίκτυο συνεργατών προσωπικού προς την Ελλάδα. Διπλασιάζουμε στην πραγματικότητα τον αριθμό των ε, υπαλλήλων που απασχολούνται στη λεγόμενη Γενική Διεύθυνση Home, δηλαδή εσωτερικών και δικαιοσύνης. Και θα ήθελα επί τη ευκαιρία να καλέσω τα κράτη-μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να ακολουθήσουν το παράδειγμα των Αυστριακών και των Γερμανών ως προς τη στελέχωση. Είδαμε κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, και εσείς και εγώ, εχθές τον Πρόεδρο Ερντογάν της ε, Τουρκικής Δημοκρατίας. η Τουρκία έχει αναλάβει ένα τεράστιο βάρος με 2,2 εκατομμύρια πρόσφυγες από το Ιράκ και τη Συρία κυρίως. Και είναι προφανές ότι χρειαζόμαστε την Τουρκία προκειμένου να προστατέψουμε τα εξωτερικά μας σύνορα. Η Επιτροπή θα πράξει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τις αξιοσημείωτες προσπάθειες της τουρκικής δημοκρατίας. Δεν μπορούμε μόνο να κοιτάμε το εσωτερικό μας, πρέπει να δούμε και την περιφέρεια της Ευρώπης για το πρόβλημα το ίδιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία λοιπόν θα πρέπει να συμπορευτούν και να αναπτύξουν αρμονικά μια πολιτική υποδοχής, προστασίας και παρακολούθησης των δύστιχων εκείνων που φτάνουν μέχρι σε εμάς. σε συμφωνία με τον ε, πρόεδρο Τούσκ και τον πρόεδρο Σούλς υπέβαλα προς εξετάσεις στον ε, Τούρκο πρόεδρο ένα σχέδιο μνημονίου για τη διαχείριση του προβλήματος των προσφύγων που θα πρέπει να συναυθεί μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 3 το απόγευμα πρόκειται να γίνει αυτή η συνομιλία. Δεν μπορώ να σας δώσω λοιπόν ακόμη απαντήσεις γιατί είπαμε ότι θα γίνει η συνομιλία στις 3 το απόγευμα με την τουρκική πλευρά η εστίαση μας όλη είναι η Ελλάδα. 66.000 πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που έχουν φτάσει στην Ελλάδα θα πρέπει να, να κατανεμηθούν σε ευρωπαϊκά κράτη. Έχω μιλήσει με την Αθήνα και το Γενικό Διευθυντή Αρμόδιο για, τη για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, κύριο Βερβέν, που από εκεί διαπραγματεύεται το πρόγραμμα που θέλω πηγηθεί για την Ελλάδα. Έχω επίση ε, συνομιλήσει και με την αντίστοιχη υπηρεσία μας στην Τουρκία την Άγκυρα για να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες της εφαρμογής ενός τέτοιου προγράμματος στην Τουρκία και έχω αναθέσει και σε πολλούς ε, αξιωματούχους μας ακόμη και στο Φραντ Τίμερμαντς που είναι δίπλα μου και δεν το ξέρει ακόμη να πάνε στην Τουρκία και να συνομιλήσουν με την τουρκική πλευρά για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας που θα συνάψουν. Αυτή η κοινή πολιτική λοιπόν μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας δεν αφορά μόνο υπαλλήλου και εξωματούχου. παρότι είναι αξιότατοι άνθρωποι. Πρέπει πιστεύω να πολιτικοποιήσουμε με την ευγενή έννοια του όρου την ε, συζήτηση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκία για το θέμα αυτό. Και οι πολιτικοί αυτοί, αυτές οι πολιτικές έχουν ένα κόστος. Παρακολουθώ. Όχι με ανησυχία, αλλά με ενδιαφέρον ένα δημόσιο διάλογο που αναπτύσσεται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή για το κατά πόσον θα πρέπει τα χρήματα τα οποία δαπανώνται από μια χώρα για τη διαχείριση του προβλήματος των προσφύγων και μεταναστών να αποκλείονται από τον υπολογισμό του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ξέρετε ότι υπάρχει μια ερμηνεία η οποία επιτρέπει να δώσουμε απαντήσεις στην υπόθεση αυτή. Δεν θέλω όμως να περάσουμε και στην απόλυτη ανευθυνότητα. Και άρα θα πρέπει, με βάση την ανάλυση στην οποία έχει ήδη την οποία ήδη έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να εξετάσουμε κατά πόσο κάποιες χώρες μπορούν να απαλλαχθούν από μια ε, υπερβολικά αυστηρή ερμηνεία του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αλλά ας μην το κάνουμε αυτό ε, ελαφρά την καρδία, γιατί αυτή τη στιγμή συζητούμε το κόστος της ανάληψης των, ε, της ευθύνης των προσφύγων. Αύριο μπορεί να υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα και η Επιτροπή είναι διαθέσιμη να συζητήσει όχι και να μπει όχι σε οποιαδήποτε περιπέτεια, αλλά πάντως να ακούσει και να συζητήσει οποιαδήποτε πρόταση. Και βεβαίως, Πρόεδρε, αφού ακούσω μεγάλη προσοχή τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα απαντήσω και στις δικές σας ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλτ Τούσκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φίλοι μου, η πραγματική δοκιμασία για οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων έρχεται σε μια στιγμή κρίσης. Όπως τις τράπεζές μας με τα τεστ κοπόσεως, Σήμερα, όπως είπε και ο κύριος Γιούγκερ, υπάρχει ένα τεράστιο τεστ ε, κοπόσεως με τους μετανάστες για να δούμε αν αντέχουν οι ομάδες των πολιτών μας. Αυτό εξέτασε το προηγούμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ξέρετε ποια ήταν τα συμπεράσματά του. Και επιτρέψτε μου να μοιραστώ κάποιες γενικότερες σκέψεις μαζί σας. Ιδίως ότι σε 10 ημέρες το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ασχοληθεί με το ίδιο ακριβώς θέμα. Οι ιστορικές αλλαγές και οι πιέσεις μεγάλης εμβέλειας απαιτούν ένα βαθμό αξιοπρέπειας και αυτοπεποίθησης από κάθε ομάδα πολιτών, ιδίως τώρα. Ολόκληρος ο κόσμος έχει στρέψει την προσοχή του στην Ευρώπη και στην αντίδρασή της στο κύμα μεταναστών που καταφτάνει. Η Ευρώπη δέχεται δρυμίες κριτικές για τις διεθνείς ε, συμβάσεις και για τη διακριτική μεταχείριση που βέβαια έρχονται να ενισχύσουν τα επιχειρήματα των ε, επικριτών μας. Και από την Ευρώπη κάποιες φωνές ε, ενώνονται με αυτά τα επικριτικά σχόλια. Όμως σε μια τέτοια προοπτική θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι η Ευρώπη είναι το χειρότερο μέρος για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες βρέθηκα απομονωμένο όταν χρειάστηκε να περασπιστώ την καλή φήμη τη Ευρώπη και να πείσω το κοινό μου ότι η αλήθεια για την Ευρώπη είναι διαφορετική στα Ηνωμένα Έθνη. Εκατοντάδε. χιλιάδε πρόσφυγε έρχονται στην Ευρώπη, διότι γνωρίζουν ότι η δική μα κοινότητα λαών είναι ακόμη η ανοιχτότερη και η πλέον ανεκτική από όλε. Εμείς σεβόμαστε τις ε, διεθνείς προδιαγραφές και συμβάσεις πάνω απ' όλα και όλοι οι άνθρωποι στην Ευρώπη είναι ασφαλέστεροι από ό,τι οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Ας μην αφήσουμε η Ευρώπη να γίνει από δύο πομπέως τράγος λόγω της ανεξέλεγκτης κριτικής μεταξύ μας. Ιδάλλως, πολύ σύντομα, οι θεοκρατίες θα αρχίσουν να μας δίνουν ε, μαθήματα για το τι σημαίνει ανοχή και ανεκτικότητα, για το τι σημαίνει δημοκρατία και όσοι είναι οι αυτούργοι για αυτή την, αυτής της τεράστιας μαζικής εξόδου θα μας ε, κρίνουν για τους πρόσφυγες. Ήδη το κάνουν. Υπάρχουν χώρες που δεν δέχονται καθόλου πρόσφυγες. Όμως, όταν θέλουν να παροτρύνουν την Ευρώπη να είναι πιο αλληλέγγυα, το κάνουν με μεγαλύτερη οξύτητα από άλλους. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προστατεύσουμε από κοινού το καλό μας όνομα. Μέλη του Κοινοβουλίου, μπορούμε να μιλάμε για αλληλεγγύη, για ποσοστώσεις και περισσότερη βοήθεια προς τους πρόσφυγες, για τις χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες, όμως να είμαστε σαφείς. Αλληλεγγύη σημαίνει αμοιβαία βοήθεια και σεβασμό. χωρί αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών δεν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε του άλλου. Είναι κοινή μα υποχρέωση να συντράβουμε του ε, πρόσφυγε και να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ταυτόχρονα. Ο καθένα θα πρέπει να φέρει πέρα σε αυτή την υποχρέωση και ταυτόχρονα Κανεί δεν θα πρέπει να εγκαταλειφθεί μόνο του να σηκώσει αυτό το βάρο. Έτσι κατανοώ εγώ την αλληλεγγύη θα πρέπει να ε, σεβαστούμε τους κοινώς επεφωνημένους κανόνες. Κάποιος είπε ότι δεν θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί το Ευρωπαϊκό Δίκαιο ή το Δουβλίνο ή οι πιστοστώσεις. Διότι έτσι θα υπονομεύαμε την έννοια της αλληλεγγύης στην κοινότητά μας. Το να σεβόμαστε τους κανόνες βέβαια σημαίνει ότι πρέπει να θυσιάσουμε και ένα μερό των συμφερόντων μας. Θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω κάποια λόγια στους Ούγγρους και Ιταλούς φίλους, τους Σλοβάκους και τους Έλληνες. Να μην έχουμε ψευδεστήσεις. Σήμερα θα πρέπει να υπολογίζουμε κυρίως στον εαυτό μας, σε εμά τους ίδιους. Κανείς δεν σκοπεύει να βοηθήσει την Ευρώπη. Που οι περισσότεροι γειτονές μας, γειτονές μας έχουν μεγαλύτερα προβλήματα να επιλύσουν και μερικοί χαίρονται με τις δυσκολίες και τα δεινά μας. Για μας οι πρόσφυγες είναι άτομα, συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι ζητούν και περιμένουν τη βοήθειά μας. Υπάρχουν βεβαίως δυνάμεις γύρω μας που θεωρούν ότι είναι μια ευκαιρία να κάνουν φτηνή πολιτική ή να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες η έλευση των προσφύγων. Είναι μια νέα μορφή πολιτικής πίεσης αυτή που ασκείται και κάποιοι το αποκαλούν έναν υβριδικό πόλεμο, μια νέα μορφή πολέμου, όπου τα κύματα αυτά ανθρώπων έχουν γίνει μια πίεση κατά των γειτόνων. Αυτό απαιτεί να επιδείξουμε ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή από πλευρά μας. Συνάδελφοι, γνωρίζετε όλοι την έννοια της ηθικής και της ευθύνης από όσα είχε πει ο Βέμπερ, ο Μάξ Βέμπερ, όχι ο Μάνφρεντ Βέμπερ. Σήμερα η ηθική και η ανάληψη ευθύνης απαιτεί να απέχουμε από ακραίες τοποθετήσεις. Και ακραίες τοποθετήσεις μιλώ και τα λόγια κατά των ε, μεταναστών από τη μία και την πρόσκληση να έρθουν όλοι όσοι το επιθυμούν, ακόμη και αν δεν μπορούμε να τους ε, πάρουμε κατά από τη στέγη μας. Πρέπει εν τέλει να καταλάβουμε το εξής. Σήμερα, πολλοί ενδυνάμοι πρόσφυγες και μετανάστες ονειρεύονται να έρθουν στην Ευρώπη. Όχι μόνο από τη Συρία, αλλά και από την Αφρική, το Πακιστάν, το Ιράκ και άλλες χώρες. Για όλους τους πρόσφυγες, η απλή εύκολη πρόσβαση στην Ευρώπη και η έλλειψη εξωτερικών συνόρων έχουν γίνει πέραν της κοινή μας πολιτικής, ένας μαγνήτης που το στραβάει προς τα εδώ, Κατά τις επισκέψεις μου στη γεωγραφική αυτή περιοχή, σε όσους μίλησα, σε μεταναστές ή πρόσφυγες, στους καταβλισμούς, στην Τουρκία ή την Αίγυπτο, όλοι μου είπαν το εξή: ότι μια ενδεχόμενη νίκη του καθεστώτος του Ασάντ πιο πιθανή σήμερα γιατί το Ιράν και η Ρωσία έχουν αναλάβει δράση στη Συρία θα οδηγούσε σε ένα τεράστιο μεταναστευτικό κύμα νέο κύμα. Χθες το μήνυμα αυτό επιβεβαιώθηκε και βάσει των τουρκικών εκτιμήσεων 3 εκατομμύρια πρόσφυγες μπορεί να έρθουν από το Αλέπ, Χαλέπι και από γειτονικά μέρη. Η αλληλεγγύη πάντοτε επικροτείται, συνάδελφοι, ενώ η ανάληψη ευθύνης και η επιμονή στην κοινή λογική. Όχι, το ίδιο. Η αλληλεγγύη όμως δεν πρέπει να μένει μόνο στα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεται και στην πράξη. Γι' αυτό ζητώ από όλους σας να αναλάβετε τις ευθύνες και να επιδείξετε κοινή λογική. Η πρώτη εντολή σήμερα είναι η αποκατάσταση του ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μια εκ των ουκάνευ προϋπόθεση για να υπάρξει αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική και πολιτική για τους πρόσφυγες. Αύριο στο Ευρωκοινοβούλιο θα ακούσατε τον Φρασουά Ουλάντ και την Άγγελα Μέρκελ. Ξέρουμε πώς εξαρτώνται από αυτή την παρέμβαση. Σε αυτή την κατάσταση της κρίσης και οι δύο έχουν δείξει την ηθική στάση τους, την οποία όλοι εκτιμούμε τα μάλα. Αύριο θα έχουμε μια ακόμη δυσκολότερη δοκιμασία. Το κατά πόσο μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη για την προστασία της ευρωπαϊκής κοινότητας και των εξωτερικών της συνόρων. Ιδάλλως και εκείνοι και όλοι μας θα είμαστε υπεύθυνοι για την ανάδυση τυχών και φραγμών στα εσωτερικά μας σύνορα. Εδώ στην Ευρώπη θα πρέπει επιτέλους να πούμε ξεκάθαρα και ηχηρά ότι η Ευρώπη χωρίς εξωτερικά σύνορα σημαίνει Ευρώπη χωρίς έγκεν. Η Ευρώπη χωρίς εξωτερικά σύνορα θα είναι ένας τόπος όπου θα καλλιεργούνται ο φόβος στον καθέναν μας. Και αυτό θα μας οδηγήσει αργά ή γρήγορα σε πολιτική καταστροφή. Τι περιμένουν οι κοινοί από τους πολιτικούς. Πάνω απ' όλα αποτελεσματικότητα και αποφασιστικότητα στις κινήσεις. Εάν υπάρχει λοιπόν μία επικρατούσα σκέψη στην πολιτική, φαίνεται αυτή τη στιγμή να μην το συνειδητοποιεί. Οι πολίτες ζητούν άλλο τρόπο να οδηγήσουμε τα πράγματα με ριζοσπαστικές λύσεις. Αυτό που θέλουν από τους πολιτικούς ευθύνοντες οι πολίτες είναι μια εγγύηση της τάξης και της ασφάλειας για την δική τους την κοινότητα. Είτε λοιπόν θα αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση ή άλλοι θα μας υποκαταστήσουν. Η πολιτική μαγιά είναι κάτι που έχει παρέλθει. Αλλά όλα θα εξαρτηθούν από τις επόμενες αποφάσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τούσκ και τώρα αρχίζει η συζήτηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κύριο Βέμπερ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Συμβουλίου για την παρουσία του εδώ. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε για άτυπο Συμβούλιο, μάλιστα, παρουσία του πρόεδρου του Συμβουλίου στη συζήτηση. Ρητά λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Αισθάνονται ανασφάλεια οι πολίτες σε σχέση με το πρόβλημα τη μετανάστευση και νομίζω ότι είναι σαφέ αυτό για όλου. και γι' αυτό θα ήθελα και εγώ από πλευρά τη ομάδα μου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, να πω στου πολίτε ότι είμαστε σε θέση να δώσουμε απαντήσει. Πριν από ένα εξάμεινο ή πριν από εννέα μήνες ποιο θα περίμενε ότι θα αναλάμβαναν δράση βρετανικά, γερμανικά, δηλαδή ευρωπαϊκά πλοία στα νερά της Ιταλίας και της Μάλτας μαζί με τις αντίστοιχες δυνάμεις. Ποιος θα έλεγε ότι θα βρίσκαμε λύσεις για 160.000 πρόσφυγες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, να υλοποιήσουμε δηλαδή την έννοια της αλληλεγγύης. Ποιος θα περίμενε στις αρχές του φθινοπόρου να δοθεί μια εντολή σαφής ε, στην Μεσόγειο για ανάληψη δράσης κατά των ε, συμμοριών των λαθροδιακινητών στη Μεσόγειο και στις ακτές Μεσογείου. Και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πως έχουμε σαφή εντολή και από τα Ηνωμένα Έθνη για να αναλάβουμε δράση και να οργανώσουμε την από εκεί προερχόμενη βοήθεια. Ε, άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να υπάρχει αμφιβολία ε, από πλευρά του πολίτη για την ικανότητα των ηγετών του να διαχειριστούν το πρόβλημα. Από την άλλη βεβαίω πολλά ζητήματα παραμένουν εκκρεμή. Από πλευρά τη ομάδα μου θα ήθελα να πω ότι δεν χρειαζόμαστε νέε ιδέε, χρειαζόμαστε υλοποίηση, εφαρμογή, εκτέλεση. Αυτή είναι η ανάγκη μα αυτή τη στιγμή. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το πακέτο μέτρων δίνει μια σωστή κατεύθυνση και σαφή βέβαια υποστήριξη έχει προσφέρει στην Επιτροπή υπό τον Ζων Κλοντ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι για την ε, προστασία των εξωτερικών συνόρων, ναι για τη διανομή, ναι για, τον, ε, για την επαναπροώθηση για τελικά τα δύο τρίτα των ε, υποτιθέμενων προσφύγων ή των ετούντων επαναπροωθούνται, ναι για την επαναπρόθεση στη χώρα προέλευσης, τρίτα κράτη ασφαλή πρέπει να προσδιοριστούν και αυτό δεν πρέπει να μείνει μόνο στα λόγια αλλά στα έργα. Ε, υλοποίηση λοιπόν, εκτέλεση, εφαρμογή απαιτείται. Και ιδιαίτερα για την Τουρκία θα ήθελα να πω δύο λόγια, μια και είχαμε χθε τη συζήτηση με τον πρόεδρο Ερντογάν. Η Τουρκία πρέπει να χαρακτηριστεί ως ασφαλές ε, κράτος προέλευσης. Υποστηρίζουμε αυτή την ε, θέση καθώς και την ε, χρηματική υποστήριξη προς την Τουρκία και την ενίσχυσή της. Αλλά θα ήθελα να καλέσω και τον Ερντογάν και την τουρκική δημοκρατία να μην λησμονούν τις αρχές γιατί το ένα κράτος είναι υποψήφιο για ένταξη πρέπει να του υπενθυμίσουμε και τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις πολιτικές αξίες και θα ήθελα να υπενθυμίσω στην τουρκική πλευρά αυτά τα, ε, αυτές τις αρχές σε σχέση με την διαμάχη της ε, στο Κουρδικό. Δεν μπορούμε να τα λησμονούμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Επίσης πρέπει να δώσουμε, και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση, προσανατολισμό στους ανθρώπους. Προσανατολισμός είναι ότι η Ευρώπη είναι η ήπειρος του ανθρωπισμού. Στο χάρτη των ανθρωπινών δικαιωμάτων καταγράφονται αυτά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τις θεμελιώδεις μας αξίες, για τις οποίες αισθανόμαστε μεγάλη περηφάνεια. Και ως εκ τούτου η Άγγελα Μέρκελ έχει δίκιο όταν λέει εμείς ως μεγάλη ήπειρος θα τα καταφέρουμε. Δεύτερον, είναι ευπρόσδεκτοι οι πρόσφυγες, αλλά ε, έχουμε και απαιτήσει. Δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα δηλαδή να ε, διεκδικήσει κανείς να πάει σε ένα συγκεκριμένο κράτος. Ε, θα πάει όπου τον στείλουν και επιπλέον έχει την υποχρέωση ο πρόσφυγας να ενσωματωθεί, να μάθει την χώρα στην οποία θα ζει, τη γλώσσα της κτλ. Και βέβαια θα πρέπει να εφαρμόζεται το κράτος δικαίου εξού και είμαι ευγνώμων ε, πρόεδρε του Συμβουλίου για το γεγονός ότι μιλήσατε για την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης, να ελέγχεται. δηλαδή ποιο μπαίνει στην Ήπειρο αυτό αλλά και ποιο επαναπροωθείται. Αυτό πρέπει και με τεχνικά, τεχνικού χαρακτήρα μέτρα να πραγματοποιηθεί ώστε να ε, υλοποιείται το κράτος δικαίου. Πρέπει να είμαστε σε θέση να ορίσουμε και ποσοστό και να κατευθύνουμε τους πρόσφυγες εκεί που πρέπει ώστε να μην χάσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών μας. Όπως έλεγα, το ΕΛΚ δεν θέλει νέες ιδέες, θέλει υλοποίηση των υφισταμένων προτάσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, το λόγο έχει ο Πρόεδρος Πιτέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο συνάδελφος έχει δίκιο. Δεν θα το περίμεναν πολύ να έχουμε τέτοια αποτελέσματα. Μεταξύ αυτών και εμείς. Εμείς στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι αυτά τα είχαμε πει ήδη από την Άνοιξη. Και καταφέραμε να τα υλοποιήσουμε τον Σεπτέμβρη. Δεν είναι και λίγο το πόσος χρόνος πέρασε. Βέβαια πρέπει να απαντούμε στις προκλήσεις αμελητή πολύ πιο γρήγορα, πρόεδρε Τούσκ. Αλλά ας προχωρήσουμε, ας προασπιστούμε αυτό τον χώρο. Εγώ θα ήθελα να είμαι Ευρωπαίος και να αισθάνομαι πρωταθλητής στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν θα ήθελα αυτή την ύπαρξη να την ε, μετατρέψω σε μια θυμωμένη και κακιασμένη αρκούδα για να αποθήσω τους ε, πρόσφυγες. Ας είμαστε λοιπόν ταχύ στις αντιδράσεις μας, ε, κύριε Τούς, με τα hot spot για, την, ε, για τον μετατόπιση, για τον συντονισμό μεταξύ της υποδοχής και της φιλοξενίας για την προστασία των εξωτερικών συνόρων, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία και το Λίβανο. Όλα αυτά με πείθουν ότι πρέπει να ε, υλοποιηθούν γρήγορα και όχι απλώς να επιρρύπτουμε ευθύνε μεταξύ χωρών χώρες που τις κατηγορούμε ενώ έχουν επομιστεί όλο αυτό το φόρτο των μεταναστών επί σειρά ετών. Ας σταματήσουμε να είμαστε αρνητικοί. Φτάνει, φτάνει να είμαστε αρνητικοί απομονώνοντας ενώ δεν μπορούμε να ε, λύσουμε τα προβλήματα. Τύχη, εγωισμοί, μίσος. Όλα αυτά αποδεικνύουν την ανικανότητα να επιλύσουμε τα προβλήματα και τα προβλήματα επιλύονται εάν είμαστε θετικοί. Ε, ας ε, σταματήσουμε λοιπόν αυτήν την στάση και ας περάσουμε σε μια νέα φάση για να μην υπονομεύσουμε το μέλλον και το πνεύμα της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πιτέλα. Εκ μέρους των συντηρητικών μεταρρυθμιστών ο κύριος Λεγκούτκο. Uh, uh Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι 800.000 μετανάστες έρχονται στην Ευρώπη. Περιμένουμε ένα εκατομμύριο, ακούσαμε από τον πρόεδρο Τούσκ. Εάν αυτά τα νούμερα ευσταθούν, είναι ξεκάθαρο ότι η ανταπόκριση την οποία έχουν σχεδιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν επαρκεί. Είναι προσεμβαλωματικές λύσεις, δεν είναι η λύση. Ως συνήθως χρησιμοποιούμε μια γλώσσα που περιπλέκει και συγχαίει τα πράγματα και την χρησιμοποιούμε για να ε, κάνουμε να σιωπήσουν αυτοί που εκφράζουν διαφορετικές απόψεις. Χρησιμοποιούμε ανθρωπιστικά επιχειρήματα, ταυτοχρόνως με τα πολιτικά επιχειρήματα. Ο, Τίμερ, ο, κ. Τίμερ μας, για παράδειγμα, έχει πει ότι η επανεγκατάσταση είναι καλή για τις ψυχές μας. Το έχετε πει αυτό, είναι τρομακτικό. Αναφερόμαστε σε εκβιασμούς. Αναφερόμαστε επίσης σε πρόσκληση προς τους μετανάστες ή τους πρόσφυγες. Η Σέγγεν έπαψε να ισχύει και μετά ε, επανα... Ε, ξαναξεκίνησε. Αυτό που θα έπρεπε να κοιτάμε όμως είναι πραγματικά ποιο είναι το μακροπρόθεσμος μας στόχος σε ποια κατάσταση θέλουμε να φτάσουμε. Έχουν αναφερθεί τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση των πολιτικών. Αυτό έχει πει το Συμβούλιο και μας φαίνεται λογικό. Όλα αυτά λοιπόν τα ταμπού, όλες αυτές οι... Ε, τα θέματα που δεν τολμούμε να συζητήσουμε στην Ευρώπη είναι το πρόβλημα. Και δεν μας επιτρέπουν να έχουμε μια λογική συζήτηση. Και αν αυτό δεν αλλάξει, τα πράγματα θα παραμένουν ίδια. Ευχαριστώ. Εκ μέρου των Φιλελευθέρων, ο σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τούσκ, ξεκάθαρα θέλω να σας πω ότι όλο και περισσότερο έχω μπουχτίσει με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όχι με σας προσωπικά φυσικά, αλλά με το θεσμικό όργανο το οποίο εκπροσωπείται. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί πρώτα απ' όλα χρειάστηκε υπερβολικά πολύ καιρό για, να για να οργανωθεί, για να συγκληθεί το έκτακτο ανεπίσημο συμβουλίο. Και δεν ήταν μια προσφυγική κρίση η οποία ξεκίνησε ξαφνικά. Αλλά εάν κοιτάξουμε και ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτού του συμβουλίου, μία σελίδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε το πιο σημαντικό, την πιο σημαντική κρίση την οποία αντιμετωπίζει την τελευταία δεκαετία η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τι κατέληξε σε μια σελίδα συμπεράσματα. και η οποία μια σελίδα εδώ που τα λέμε απλώς επαναλαμβάνει ε, αποφάσεις οι οποίες είχαν ήδη ληφθεί από τους Υπουργούς Εσωτερικών για τον αριθμό των προσφύγων οι οποίοι θα μετεγκατασταθούν και κάποια κονδύλια. Και αναρωτιέμαι αγαπητοί συνάδελφοι, οι άνθρωποι από τη Συρία, πόσοι ακόμα μάλλον άνθρωποι από την Συρία πρέπει να προσπαθήσουν να φτάσουν στην Ευρώπη και να πεθάνουν στο δρόμο πριν να αποφασίσει το Συμβουλίο ότι χρειάζεται να αναλάβει μια συνολική, συνεκτική δράση επί του θέματος, όπως εξάλλου έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι και κάτι καινούριο. Έχετε προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας έχει προτείνει ένα συνεκτικό και συνολικό σχέδιο το οποίο συμπεριλαμβάνει ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου το οποίο θα ξεπεράσει τις προβλέψεις του Δουβλίνου. Ένα νέο σύστημα για την μετανάστευση, ε, το οποίο θα ενοποιήσει τα συστήματα ε, τα μεταναστευτικά στην Ευρώπη. Αντί για να έχουμε 28, μια κοινή ε, πολιτική για την μπλε κάρτα, μια κοινή πολιτική για την φύλαξη των συνόρων, των χερσαίων και των θαλασσίων. Όλα αυτά λοιπόν έχουν τεθεί στο τραπέζι, αλλά στις 11 Σεπτεμβρίου αρνήθηκε το Συμβούλιο να τα συμπεριλάβει στα συμπεράσματα του. Δεν τα έχει συζητήσει. Λοιπόν, αναρωτιέμαι τι χρειάζεται πια να γίνει για να αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αναλάβει τις ευθύνες του, να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις πάνω στο πακέτο που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. όπως εξάλλου έχει ήδη τοποθετηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάνω σε αυτά τα θέματα. Και αναρωτιέμαι γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Γιατί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν καταφέρνει να ξεπεράσει ε, τα εσωτερικά του προβλήματα και η απόψη μου ε, ε, είναι ξεκάθαρη. Εγώ θα ήθελα το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να συμφωνήσουν να δώσουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να προχωρήσει γρήγορα με fast track διαδικασία στις προτάσει τη. Όσον αφορά τώρα τα εξωτερικά σύνορα, δεν έχει έρθει άραγε η στιγμή ακόμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνολικά η κυρία Μογκερίνη, το Συμβούλιο, όλοι να λάβουν πρωτοβουλία όσον αφορά την σύγκρουση στη Συρία. Το μόνο που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να ενισχύουμε ε, βομβαρδισμούς, βομβαρδισμούς αμάχων στη Συρία. Και ε, σε αυτούς τους βομβαρδισμούς τώρα προσθέθηκαν και οι βομβαρδισμοί των Ρώσων ε, που σκοτώνουν αμάχων. Δεν κοιτάμε λοιπόν ποια είναι τα γενεσιουργά αίτια αυτών των ε, ε, προσφυγικών ροών. Οι Αμερικάνοι ξεκίνησαν την επέμβαση στην Συρία. Τι κάνει η Ευρώπη, απλώς δέχεται τους πρόσφυγες που προσκλήθηκαν από αυτήν. Και δεν συζητούμε καν για το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής. Ε, θα πρέπει λοιπόν να αναλάβετε πρωτοβουλία. θα πρέπει να δώσετε εντολή στην κυρία Μογκερίνη να, να, να, να δραστηριοποιηθεί. Επίσης όσον αφορά το τις ε, ζώνες ε, αεροπορικού αποκλεισμού. Έχει τεθεί το θέμα και ακούω ότι χρειάζεται εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μα για να βομβαρδίζουμε Σύριους αμάχους δεν χρειαζόμαστε εντολή από τον ΟΗΕ, για να επιβάλλουμε αεροπορικό αποκλεισμό χρειαζόμαστε. Επίση, τίθεται το ζήτημα τη χρηματοδότηση. Πρέπει να ε, εξευρεθούν δωρητέ, κράτη δωρητέ. Εσείς κύριε Τούσκ ε, εκπροσωπείτε μια ολόκληρη ήπειρο, όχι απλώ μια χώρα. Πρέπει να αναλάβετε τι ευθύνε σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριο εκ μέρου τη ΓΚΟΕ. Μάλιστα, δεν είναι εδώ. Καλώς. Σας παρακαλώ. Ποιος θέλει το λόγο. Μπλάνκο νόμιζα ότι σας λέγανε. Κύριε Μπλάνκο, παρακαλώ εσείς. Πρόεδρε, η υποχρέωση ενός βουλευτή είναι να βρίσκεται μέσα στην ε, Ολομέλεια για να συμμετέχει στη συζήτηση. Λυπούμε που, εδώ, που δεν είναι εδώ ο κύριος ε, Ιγλέσιας. Εντάξει, ναι, αλλά μπορεί και να έρθει αργότερα, λέει ο πρόεδρος. Πράσινη, Λάμπερτς. Κύριε Πρόεδρε, τους σας άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Νομίζω ότι ω Ευρωπαίοι πρέπει να παραμείνουμε υπερήφανοι για όσα έχουμε καταφέρει και οικοδομήσει στην Ευρώπη. Έχετε δίκιο. Και είναι αλήθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι άψογη. Το κράτο δικαίου ακόμα βρίσκεται υπό οικοδόμηση. Οι δημοκρατίε μα κάποιε φορέ δεν στέκονται απόλυτα στο ύψο του. Όμω, ακόμα και αν υπάρχουν αυτέ οι ατέλειε, και πάλι εδώ θα διάλεγα να ζήσω χωρί δισταγμό. Και αυτό πιστεύουν και πολλοί μετανάστε, πρόσφυγε ή ετώντε άσυλο που θέλουν να έχουν πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε δίκιο που λέτε ότι μα δίνουν μαθήματα θρησκευτική ε, ανοχή ή δημοκρατία ή θεοκρατία. Είναι κάπω ε, θρασί. Το λιγότερο μπορεί να πει κανεί. Κύριε Τούσκο, όμω, οι χώρε στι οποίε επενήσεστε όταν το λέτε αυτό, συνήθω είναι σύμμαχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να σας ακούσω να απευθύνεστε σε αυτά τα κράτη και να τους λέτε όσα μας είπατε. Θα ήθελα όταν είδατε χθε τον κύριο Ερντογκάν και τη στιγμή που καταπιέζει τον τύπο ή τη δικαιοσύνη στη χώρα του, ξαναξεκινάει τον πόλεμο στη δική του χώρα, εκεί πώς μπορούμε να ενώνουμε τις δυνάμεις μας ε, μαζί του. Είναι σαν να μην υπάρχει τότε αυτό το θέμα. Θα ήθελα λοιπόν εκεί να, να δείχνετε κάποια ταπεινοφροσύνη, αν και έχετε δίκιο. Πρέπει να είμαστε περήφανοι που είμαστε Ευρωπαίοι. Επίση, είπατε ότι πρέπει να αποφύγουμε τι ακραίε τοποθετήσει. Και πάλι θα συμφωνήσω μαζί σα. Αλλά να σα δώσω δύο αριθμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει το 23,7% του ε, διεθνούς ΑΕΠ, δηλαδή του διεθνού πλούτου. Και με τι 60.000 πρόσφυγε που πρέπει να κατανεμηθούν στην Ευρώπη έχουμε να αντιμετωπίσουμε 0,2% των προσφύγων στον κόσμο ολόκληρο. Εάν λοιπόν έχουμε φτάσει κοντά σε μια ακραία τοποθέτηση, δεν έχουμε φτάσει σε καμία περίπτωση στο άκρο του να ανοίξουμε τις πόρτες μας ορθάνυχτες. Θα μπορούσε λοιπόν να τα πάει καλύτερα σε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα σας παρακαλέσω να ακολουθήσετε τις ε, παροτρύνσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακούσαμε επανειλημμένω εδώ τον κύριο Γιόνκια και τον κύριο Τιμερμανή να σα ζητούν να ζητήσετε από τα κράτη-μέλη να προβλέψουν μια κλίδα κατανομή των προσφύγων μόνιμη. Του άκουσα τους ίδιους να σας ζητούν να προβλέψετε νόμιμες οδούς πρόσβασης ε, στην Ευρώπη για να πάψουν οι θανατηφόρες ε, μεταβάσεις μέσω των εμπόρων. Και επίσης σας ζήτησα να ιδρύσετε μια ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου. Εδώ υπάρχουν ακόμη πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν. Κάποια βήματα έγιναν κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά είναι απλώς μια αρχή. Συνεχίστε τον ίδιο αγώνα. Ευχαριστώ. die EFDD-Fraktion spricht jetzt Herr Κύριος Καστάλντο, Ευρώπη των Ελευθερών και των Δημοκρατιών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ειλικρινά, έχοντας ακούσει τα σχόλια αυτού του άτυπου συμβουλίου, παραμένω άναυδος. Κάποιοι χαίρονται με τα αποτελέσματα τα οποία επιτέχθηκαν. Δεν ξέρω σε ποιο κόσμο ζουν. Στον, στην κρίση αυτή των προσφύγων με βουνά νεκρώνεται να έχουμε κάνει ένα πολύ μικρό βήμα. 100.000 ε, μετανάστες έρχονται ακόμη προς την κατεύθυνσή μας. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια κρίση τυφλότητας της Ευρώπης, όπου κάποιοι κοιτούν από την άλλη, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άτομα έρχονται στην επικρατειά μας και τους αποθούν να φύγουν ως το δυνατόν πιο γρήγορα. Κάποιοι καταγράφουν, κάποιοι άλλοι χρησιμοποιούν τα σειρματοπλέγματα και τα δακρυγόνα ή την ε, πραγματική σωματική βία. Εδώ μιλάμε για μια κρίση όχι των εξωτερικών μα συνόρων, κυρίε και κύριοι, αλλά των εσωτερικών σύνορων. Ένα τείχο ε, στη Βουδαπέστη ε, χωρίζει τη χώρα. Αν η Βουδαπέστη αποφασίζει ένα τείχο να τη χωρίζει από τη Σλοβενία, που είναι και αυτό μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό σημαίνει ότι κράτη όπω η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Ουγγαρία έχουν περάσει ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Θυσιάζοντα ε, τι κοινέ μα αξίε, τα εκλογικά συμφέροντα κάποιων. Η συνεργασία με την Τουρκία είναι κάτι που το γιορτάζουμε, ενώ ξεχνάμε το πώ υποφέρει ο κουρδικό λαό. Έτσι χάνουμε την αξιοπιστία μα και αυτή είναι η Ευρώπη σήμερα. Δεν είναι η Ευρώπη του κάνουμε βήμα από το βήμα πρόοδου, αλλά χτίζουμε τείχο μετά το τείχο. Α φροντίσουμε λοιπόν να λάβουμε ανθρωπιστικά μέτρα, πραγματικά μέτρα, να έχουμε νόμιμε οδού πρόσβαση, να ξεπεράσουμε το Δουβλίνο όπω είναι σήμερα ή τι εμπορικέ πολιτικέ ε, εκμετάλλευση ή τα όσα δεν κάνουμε για τι κλιματικέ αλλαγέ. Φτάνουν τα μικρά βήματα, χρειάζονται θαραλέα άλματα. Αυτέ είναι οι επιλογέ που πρέπει να κάνουμε και αυτέ είναι που θα μα δώσουν καλό όνομα, κύριε Τούσκ. Εμεί μπορούμε. Εσεί πότε, εάν όχι τώρα. E η από την ομάδα ΙΕΝΕΦ, e η κυρία Αλιού. Ο κύριος Αλιού. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Χρειάστηκε να περάσουν πολλές εβδομάδες και να δούμε μια φρικτή ε, φωτογραφία για να φτάσουμε να πούμε το όρος Ευρώπη έτε και μην. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν τη βοήθεια, ναι, στα κράτη που αντιμετωπίζουν ε, τα προβλήματα στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, τους φίλους από την Ιταλία και την Ουγγαρία. Αλλά σταματήστε να στιγματίζετε την Ουγγαρία του κυρίου Ορμπάν που σε κατάσταση κατεπίγουσα χρειάστηκε να ε, δράση για να αντιμετωπίσει αυτό το χάο μέσα από την κακοφωνία που έβγαινε από το Συμβούλιο. Θα σα θυμίσω ότι το 1956 η Αυστρία είχε μέσα σε μερικέ εβδομάδε δεχθεί 170.000 πρόσφυγε που έφευγαν κυνηγημένοι από τον κομμουνισμό. Η Ευρώπη των 28 δεν είναι σε θέση να λάβει την ελάχιστη απόφαση. Πώ λοιπόν να μην δούμε ότι σήμερα υφιστάμεθα τι συνέπειε των δικών σα σφαλμάτων του παρελθόντο την ε, προσχώρησα στην τυφλή, στην ε, νέα παγκόσμια τάξη του Μπούς με τους πολέμους στο Ιράκ, την Συρία, την ε, Λιβύη, την Αίγυπτο με αθώα θύματα, με θύματα καθημερινά. Δεν λειτουργούν λοιπόν τα συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι, παρα, είναι παραλυτό αυτό το σύστημα, βρίσκεται σε μια κατάσταση σκλήρινσης και όπω έλεγε ο στρατηγός Δεγκόλ, πρέπει να δείξετε εμπιστοσύνη στα έθνη και στην εθνική κυριαρχία και θα δείτε τότε ότι η αποτελεσματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη. Ο κύριος Παπαδάκης, μία βουλευτής. Το μικρόφωνο σας κύριε Παπαδάκη με τις αποφάσεις της συνόδου η ευρωπαϊκή ένωση διατηρεί το μεγάλο όγκο προσφύγων και μεταναστών στην κόλαση των υπεριαλιστικών πολέμων τη φωτιά των οποίων άναψαν η ίδια και οι σύμμαχοί της το νατο η ευρωπαϊκή ένωση και οι άλλοι υπεριαλιστές με τους ανταγωνισμούς τους για τα συμφέροντα των μονοπωλίων. όσο για τους πρόσφυγες που από τα νύχια των κυκλωμάτων φτάνουν στα κέντρα επιλογής hot spots τους κοιτούν στα δόντια και επιλέγονται μόνο οι απαραίτητοι για την καπιταλιστική αγορά εργασίας για τους υπόλοιπους τους περισσότερους η ευρωπαϊκή ένωση και οι κυβερνήσεις της αποφάσισαν καταστολή και απελάσεις. όσο για τον κανονισμό του δουβλίνου και τους άλλους μηχανισμούς καταστολής της ευρωπαϊκής ένωσης τις δυνάμεις ταχείας επέμβασης αυτοί ζουν βασιλεύουν και ενισχύονται και οδηγούν σε νέες εκατόμβες νεκρών μετατρέπουν σε σταθμό συγκέντρωσης προσφύγων την ελλάδα το κκε καλεί το λαό το εργατικό λαϊκό κίνημα να δυναμώσει την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες ενάντια στην πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης και να διεκδικήσει ανάμεσα σε άλλα την απευθείας μεταφορά τους από τα σημεία εισόδου στις χώρες τελικού προορισμού τους με δαπάνες της ευρωπαϊκής ένωσης και το οηε. Ο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Πρόεδρε, τα μαζικές κινήσεις προσφύγων και μεταναστατών θα είναι η μεγάλη πρόκληση της επόμενης 20 Θα πρέπει να δώσουμε ένα σύστημα λοιπόν το οποίο να εξασφαλίζει και την νόμιμη μετανάστευση προς την Ευρώπη και να δίνει απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα προβλέποντας ότι δεν ε, ε, καταργούνται τα εξωτερικά σύνορα. Ταυτόχρονα χρειάζεται ελληνική μεταξύ των κρατών, να εξασφαλιστεί δηλαδή η συνεργασία με τις χώρες της διέλευσης ε, όπως η Τουρκία που θα εξασφαλίσει διασφαλίζουν ότι όποιος μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπαίνει νόμιμα και ε, αυτοί που χρειάζονται βοήθεια θα την λαμβάνουν ώστε να εξασφαλίσετε για όλους η ασφάλεια και η προστασία. Ένα κοινό μέλλον λοιπόν το απαιτεί αυτό γιατί δεν υπάρχει μόνο η Συρία. Μετά τη Συρία υπάρχουν και άλλοι πολλοί μετανάστες και πρόσφυγες από πολλές άλλες χώρες. Πρόεδρε, πλησιάζει ο χειμώνα, όπως έλεγε και τις προάλλες στην Ολομέλεια ο κύριος Τούσκ. Πλησιάζει ο χειμώνα, πολλοί δρόμοι κλείνουν θα είναι λιγότεροι αυτοί που θα φτάνουν γιατί δεν θα μπορούν να διασχίσουν τις θάλασσες και θα τους χάσουμε από τις οθόνες της τηλεόρασης, θα τους λησμονήσει ο κόσμος γιατί ό,τι δεν περνάει στην τηλεόραση είναι σαν να μην υπάρχει. Σφάλμα τεράστιο θα διαπράταμε λοιπόν αν το πράξουμε αυτό και αν αναβάλαμε για περισσότερο το πρόβλημα διότι θα χειροτερεύσει ακόμα την προσεχή άνοιξη. Υπάρχουν μέτρα κύριε Τούσκ, φροντίστε να τα σεβαστούν τα κράτη-μέλη. Αν ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε πρέπει πια να πάψουμε να μιλάμε και να αρχίσουμε να πράττουμε. Ο πρόεδρος Σοσιαλιστές Δημοκράτης, κυρία Φαϊόν. Ευχαριστώ. Χρειάστηκε εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες να φτάσουν στην Ευρώπη για να ξεκινήσουμε να αναλαμβάνουμε δράση. Τα μέτρα για την επανεκατάσταση που αποφασίστηκαν είναι ένα θετικό βήμα, αλλά η κατάσταση όπως έχει σήμερα μας δοκιμάζει όλους, δοκιμάζει την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επίσης και το μέλλον της, τις νέες κατευθύνσεις που θα χρειαστεί να ε, πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να παραμείνει ένας ε, χώρος ε, ανταγωνιστικός και ευημερών. Σύντομα θα δούμε ποια είναι αυτά τα κράτη-μέλη που θα αναλάβουν τα βάρη που τους αναλογούν, ποια είναι αυτά τα κράτη-μέλη τα οποία επιδιώκουν να ε, ε, σεβαστούν τις αρχές της ελληνικής και ποια είναι εκείνα τα οποία απλώς προσπαθούν ε, να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Να αναφερθώ στην Σλοβενία. Η Σλοβενία έχει παράσχει βοήθεια στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Πολλέ αλλαγέ θα συμβούν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο τα επόμενα χρόνια, αλλά οι μετανάστες μπορούν να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις που θα εμφανιστούν, για παράδειγμα τις δημογραφικές προκλήσεις. Δεν θέλουμε να ξαναορθώσουμε τύχη ανάμεσα στις ε, χώρες ε, της Υπήρου μας. Δεν θέλουμε στη Σλοβενία να ξαναδούμε ε, έναν φράχτη να, χωρίζει, να μας χωρίζει από τους γείτονες μας Ούγκρους. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους να συνεννοηθούμε. Δεν χρειαζόμαστε να ρίξουμε λάδι στη φωτιά σε εντάσεις που υπάρχουν στα Δυτικά Βαλκάνια, όπως ε, διαπιστώσαμε να συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες. Αν ακολουθήσουμε ένα τέτοιο δρόμο θα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Φαγιώνο. Ο κύριος Τσίλεκ, μέρους ομάδας συντηρητικών μεταρρυθμών. Μισθών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ευχαριστούμε για αυτή την ανοιχτόμυαλη τοποθέτηση και την ε, ε, παρατήρηση για, τις, για τον νέο υβριδικό πόλεμο και το πόσο τρίτες χώρες ε, μπορεί να μεταλλεύονται την ευκαιρία για να ασκούν πίσω στα εξωτερικά σύνορα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την κατανομή που προτείνει τις υποχρεωτικές ποσοστώσεις προκαλεί μια καχυποψία των πολιτών έναντι των ευρωπαϊκών, θεσμών και υπάρχουν διχασμοί εντός της κοινωνίας. Κανείς δεν μένει αδιάφορος στο πρόβλημα των προσφύγων. Δεν θέλουμε όμως να υπάρξει και κριτική μεταχείριση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω διαχείρισης από μέρος μας. Θα ήθελα λοιπόν μια απάντηση από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πώς θα μπορούσαμε να βρούμε μια δημοκρατική απάντηση, γρήγορη απόκριση και στα θέματα που αφορούν την κατάσταση της, στην Καταλωνία. Ποια θα ήταν η απόκραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλημέρα σε όλους, να συνεχίσουμε τη συζήτηση και τώρα η κυρία Κέλλερ για ένα λεπτό. Παρακαλώ. Ναι, πρέπει να μιλήσουμε για τις επιτυχίες πολύ καλά, αλλά να κοιτάξουμε και την πραγματικότητα 160.000 πρόσφυγες που έχουν φύγει από τις αιστείες τους και Ακόμα δεν έχουμε τους 8.000 ε, χρόνια τώρα ζητάει περισσότερα χρήματα η πατιαρμοστία για τους πρόσφυγες και όμως ακόμα δεν έχουν ε, διατεθεί. Πού βρίσκεται η απόφαση του Συμβουλίου προκειμένου να εξασφαλιστούν επιτέλους νόμιμες ε, μέθοδοι, νόμιμες διαδικασίες για μετανάστευση για να μην τους ρίχνουμε στα χέρια των λαθροδιακινητών τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό το παλιό σύστημα του Σέγγεν το πεπαλαιωμένο και πρέπει πλέον να πούμε ότι προτιμούμε, να ομολογήσουμε ότι προτιμούμε να αφήσουμε το πρόβλημα να το επιλύσουν άλλα κράτη έξω από εμά. Αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο σύμφωνο. Η συμφωνία με την Τουρκία δηλαδή. Φαίνεται δηλαδή να έχουμε πει στον Ερντοάν, κοιτάξτε, κρατήστε του εσεί και εμεί θα σταματήσουμε να σα επικρίνουμε για το κουρδικό, για την ελευθερία του τύπου και για τα λοιπά προβλήματα. Κύριε Τούσκ, δεν είναι αυτή η Ευρώπη για την οποία μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πάξας για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η στήριξη με δισεκατομμύρια ευρώ θα επιλύσει την κρίση αυτών των προσφύγων. Όχι, διότι οι πολίτε στην Ευρώπη δεν βλέπουν χειροπιαστά αποτελέσματα που θα του έδιναν ελπίδε. Ποια είναι τα γενεσιουργά αίτια του όλου φαινομένου. Όταν αντιμετωπίζουμε απλώ τα συμπτώματα, το σύστημα επανεγκατάστασης των προσφύγων δεν αρκεί. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να ε, ελέγχουμε και να προστατεύουμε καλύτερα τα εξωτερικά μας σύνορα. Υπάρχουν χώρες που προσπαθούν να προστατεύουν τα εξωτερικά τους σύνορα, αλλά αποκαλούνται εχθροί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό αποτελεί άμεση παρέμβαση στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία τους. Η έλευση των προσφύγων είναι απλώς το προανάκουσμα μιας μελλοντική κρίσης. Πρέπει να έχουμε ισχυρές αρχές για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας. Δεν χρωστάμε τίποτα σε κανέναν. Ε, θέλουμε να δεχτούμε ε, τους πετσεκλημένους μας, αλλά αυτούς που θέλουν να μπουν με το ζόρι από την πόρτα, από το παράθυρο, πρέπει να τους αποθήσουμε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πάσκας έχει μια γαλάζια κάρτα από τον κύριο Κόμπορν. Παρακαλώ, κύριε Κόμπορν. Πρόεδρε, εγώ διαπιστώνω με αυτή τη ε, συνεδρία του Συμβουλίου ότι έχουμε αποτύχει πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε μπορέσαμε να δώσουμε απαντήσεις ε, στο οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας, ούτε τώρα μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις στο προσφυγικό. Και ε, βλέπουμε ότι ολόκληρη η Ευρώπη αποδεικνύεται ανίκανη να λάβει αποφάσεις. Ρωτώ, λοιπόν Κάποιοι λένε α, θα τους κάνουμε δεχτού όλους τους πρόσφυγες. Ε, όχι, αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει χιλιάδες ε, χιλιόμετρα δρόμου, αλλά θα τους δεχθούμε όλους. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μία λύση εφόσον τα κράτη επανέρχονται και διεκδικούν και πάλι την εθνική τους κυριαρχία για να λαμβάνουν εκείνα τις αποφάσεις. Και έχουμε έρθει πλέον σε μία κατάσταση όπου βρισκόμαστε σε μία κατάσταση ε, εκβιασμού σε σχέση με τους Τούρκους, με τους Τούρκους επαναλαμβάνω, και δεν είμαστε σε θέση να ε, δώσουμε απαντήσει στα προβλήματα. Θα πρέπει βεβαίως να καταπολεμήσουμε πολεμηθεί το Ισλαμικό κράτος και χαιρετίζω το, τις προσπάθειες των Ρώσων μαζί με τους Αμερικανούς. Τώρα μόνο οι Ρώσοι, οι Ρώσοι το πράττουν, δηλαδή να καταπολεμηθεί το Ισλαμικό κράτος, να εξασφαλιστούν ασφαλείς ζώνες και στα αραβικά κράτη και στα νησιά της Μεσογείου έτσι ώστε να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι και να υπάρξουν περιοχές προστασίας για τους ανθρώπους αυτούς. Υπάρχουν λύσει, μόνο που δεν τις θέλουν οι σοσιαλιστές και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκόλνη, ένα λεπτό, έχετε το λόγο. Στις 23 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, το αποφάσισε το Συμβούλιο ότι θα προσκαλέσουμε 800.000 ε, μετανάστες και πολιτικούς πρόσφυγες, αλλά γνωρίζουμε ότι η συντριπτική τους πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων δεν είναι πολιτικοί πρόσφυγες. Γιατί, λοιπόν, δεν μιλούμε ξεκάθαρα για τους αυτούς που είναι πραγματικά πολιτικοί πρόσφυγες, αυτούς που πραγματικά χρειάζονται διεθνή προστασία, που θα έπρεπε τους δύο του Τζούλια Νασάνς για παράδειγμα και του, τον Σνόντεν τους δύο πραγματικούς πολιτικούς πρόσφυγες πρέπει να έχει προστατεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο δεν τα κατάφερε και είναι για, τα, για τη θεσμική της ε, δομή αυτό. Το 2013 προσπάθησε από την Ιταλία, από τη Γαλλία ε, να ζητήσει πολιτικό άσυλο και αυτές οι χώρες έκλειναν τα σύνορά τους, τον εναερίο τους χώρο. Ο Ασάνς βρέθηκε εγκλωβισμένος στο, στην πρεσβεία του Εκουαδόρ στο Λονδίνο. Έξι εκατομμύρια λίρες έχει κοστίσει αυτή η ιστορία στους ε, Βρετανούς ελευθερία στον Ασάνς, ελευθερία στον Σνόντεν. Ευχαριστούμε κύριο Σκόρμπιχτ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια τεράστια πρόκληση εδώ στην Ευρώπη. Αυτά που είπατε και ο τρόπος που τα παρουσιάζετε, το περιεχόμενο της παρουσίασής σας, δεν αντιστοιχούν στη βαρύτητα του θέματος και τη σοβαρότητά του. Εμείς κατανοούμε ότι το πρόβλημα είναι οι εντάσεις εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Υπάρχει ανάγκη κάτι να αλλάξει, να αλλάξει κάτι στον τρόπο που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τόνος της παρουσίασής σας δείχνει ε, με τη δραματικότητά του ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Η έκκληση μου κύριε Τούσκ ε, είναι η εξή. Ποια είναι η άποψή σας για την κατανομή των αρμοδιοτήτων. Τι θα έπρεπε να κάνουν τα κρατημέλη μαζί και τι ξεχωριστά για το θέμα αυτό. Και ποια είναι εδώ η αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι αποφάσεις που λαμβάνει συνάδουν με τη συνθήκη. Μιλάμε για ένα χρονικό σημείο όπου καλό θα ήταν να πανεξετάσουμε το όσα κάνουμε. Διότι η κατάσταση, όπως είπατε και εσείς, είναι δυσχερέστατη. Ευχαριστούμε, κύριε Όλμπριχτ. Ε, έχετε μια γαλάζια κάρτα από τον κύριο Έτβικ. Παρακαλώ. Όχι, ο κύριος Έτβικ. No, Un momento. Μισό λεπτό. Κύριε Έτβικ, παρακαλώ. Thank you. You can see how keen we are on this. Πρόεδρε, βλέπετε πόσο μας αρέσει να κάνουμε ερωτήσεις στους συναδέλφους και η ερώτησή μου είναι πολύ απλή. Μπορείτε να με βοηθήσετε να αντιληφθώ ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που μιλάνε σήμερα τι έχει γίνει. Όλοι λέτε αλλαγή, εξωτερικά σύνορα, να μην μας κατακλείσουν όλοι αυτοί. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που τα λένε αυτά. Δεν είναι αυτοί οι οποίοι αναφανδόν ψήφιζαν υπέρ των πάντων, να δεχθούμε να έρθουν και περισσότεροι, να ενθαρρύνουμε τα ρεύματα. Μπορείτε να με βοηθήσετε να καταλάβω ποιο μιλάει επιτέλους σήμερα. Δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Κύριε Όλμπριχτ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ας κάνω μια επαλήθευση αν θέλετε. Εγώ θα μπορούσα να σας δώσω μια απλή απάντηση. Εάν κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα φραγμό, ας κάνουμε μια επαλήθευση να δούμε ποιο είναι πραγματικός πρόσφυγας. Και τότε αν είναι να του στείλουμε στα σπίτια τους. Ο κύριος Γκερέρο, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Την προηγούμενη εβδομάδα επισκέφθηκα τον Λίβανο και την Ιορδανία με αντιπροσωπεία της πολιτικής μου ομάδας ως μόνιμος εισηγητής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανθρωπιστική δράση. Εκεί είδαμε εκπροσώπους των ε, Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, για την Παλαιστίνη, ε, από την UNICEF, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εκπροσώπους κάποιων εκ των αρχών των χωρών αυτών, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, παραδείγματι επισκεφθήκαμε τα, τους καταβλισμούς προσφύγων του Μπαχάρη και του Μάχη Μπαχανέ στο Λίβανο. Δύο καταβλισμούς λοιπόν που υποδέχονται 120.000 πρόσφυγες. Ο ένας βρίσκεται στον Λίβανο, ο άλλος στην Ιορδανία. 120.000, τον ίδιο ακριβώς αριθμό που συζητούμε αν θα δεχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σύνολο των ε, συστάσεων που ακούσαμε στις συναντήσεις αυτές λοιπόν ήταν συνοπτικά το εξής. Η Ευρώπη να δουλέψει ενωμένη για να βρει μια λύση στον πόλεμο στη Συρία γιατί αν ο πόλεμος της Συρίας ε, αγγίξει τη Δαμασκό αν φτάσει στη Δαμασκό, αν επικρατήσει αυτό το κράτος, το λεγόμενο Ισλαμικό, τότε θα είναι εκατομμύρια οι πρόσφυγες οι οποίοι θα πάρουν το δρόμο και θα πνίγονται για να φτάσουν σε ακτές της Μεσογείου. Αυτά μας είπαν. Μας είπαν ότι πρέπει να διατηρήσουμε την, και να συντηρήσουμε την ελληνική με τον Λίβανο και την Ιορδανία, γιατί αν καταρρεύσουν τα κράτη αυτά, εκατομμύρια πρόσφυγες από τους δικούς τους καταβλισμούς θα πάρουν το δρόμο. Πρέπει να αποφύγουμε δε και μία τρίτη τυφάδα, για την οποία πολλής λόγος γίνεται αυτό το καιρό. Πρέπει να επιδείξουμε αποτελεσματικά αλληλεγγύη. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να επιδείξουν αλληλεγγύη. Πρέπει να προσφέρουμε δε την παιδεία στα παιδιά, την εκπαίδευση στα παιδιά που βρίσκονται στους γιατί αν δεν έχουν τα παιδιά αυτά ευκαιρία να, στελούν, να πάνε στο σχολείο, θα πάρουν το δρόμο αναγκαστικά οι γονείς τους της προσφυγιάς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόμπουρν έχει μια μπλε κάρτα για σας, κύριε Γκερέρο, τη δέχεστε. Micro. Does that? Ε, Συμφωνείτε μαζί μου κύριε Κεραίρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να στέλνει από εδώ και από εκεί στις διάφορες χώρες της Ευρώπης τους ανθρώπους θα μπορούσε καλύτερα να επευθυνθεί στο Κουβέιτ και στη Σαουδική Αραβία για να χτίσουν προσφυγικούς καταφυλισμούς στα σύνορα αυτών των χωρών με τη Συρία. Δεν θα ήταν αυτό μια πολύ καλύτερη πολιτική από το να μετακαθιστούμε ανθρώπους από εδώ και από εκεί στην Ευρώπη. Συμφωνείτε μαζί μου κύριε συνάδελφε. Κύριε Κόμπουρν, λίγα πράγματα μπορώ να φανταστώ ότι θα κατέληγα σε συμφωνία μαζί σας, σε λίγα πράγματα θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά το θέμα είναι να κοιτάξουμε εμείς τι οφείλουμε να πράξουμε, όχι άλλοι. Γιατί εμείς έχουμε ευθύνες. Η υπευθυνότητα να δώσουμε απαντήσεις είναι δική μας πρώτα απ' όλα. Μετά θα ζητήσουμε από τους άλλους να βοηθήσουν και αυτοί. Ευχαριστώ, επόμενος ομιλητής, η κυρία Τρεμπέσιους. Ένα κύμα μεταναστευτικό κατακλείζει την Ευρώπη. 1,5 εκατομμύρια αναμένεται να φτάσουν έως τη Γερμανία εφέτος και αυτό βέβαια εξωτερώνει αδίποτε μέχρι τώρα πρόβλεψη. Η κατάσταση έχει βγει εκτό ελέγχου στο Συμβούλιο των Υπουργών των, ε, στη Σύνοδο Κορυφή. Έγινε λόγος για 160.000 ε, ή 180.000 μετανάστες που θα έφθαναν ε, και θα κατανέμονταν μεταξύ των κρατών της Ευρώπης. Αλλά προφανώς έχει χαθεί κάθε έννοια πραγματικότητας και ε, σχέση με την πραγματικότητα από την ε, καγκελάριο της Γερμανίας εάν δεν αναγνωρίζει ότι πρόκειται να φτάσουν πολύ περισσότεροι και δεν μπορούμε να αφήσουμε τους ε, δήμους και τις κοινότητε να διαχειριστούν τα προβλήματα αυτά. Πρέπει να κλείσουμε τα σύνορα και πρέπει να αποστείλουμε σαφή μηνύματα προς τους μετανάστες ότι η Ευρώπη δεν είναι σε θέση να του κάνει όλου δεκτού. Σήμερα οι περισσότεροι πρόσφυγες βρίσκονται υπό την ε, προστασία και διαχείριση της ΥΠΑ της των Ηνωμένων Εθνών μέσα στην Ευρώπη. Πρέπει να καταστήσουμε σαφές λοιπόν ότι δεν μπορούν να έρχονται στην Ευρώπη, είναι ασφαλείς εκεί που βρίσκονται και δεν χρειάζεται να φτάνουν μέχρι την Ευρώπη. Κυρία Τρεμπέζιους, έχετε μπλε κάρτα και υπενθυμίζω στους συναδέλφους ότι μπορούμε να κάνουμε δεκτή μόνο μία μπλε κάρτα για κάθε βουλευτή. Είχε ζητήσει το λόγο λοιπόν ο κύριος Κέικ που έχει στήσει το λόγο. Γκέριγκερ. όχι, δεν είχατε στήσει εσείς μπλε κάρτα. Γιάκον Σάρι. Te puhuitte luon, ikään kuin luonnonvoimista Κύριε Πρόεδρε, μιλούμε για προσφυγικά κύματα, για ροές, ενώ στην πραγματικότητα αναφερόμαστε σε ανθρώπους. Και αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε να καταλάβουμε ποια είναι η κατάσταση, να την αντιμετωπίσουμε στο σύνολό τη, να βρούμε ε, θέσεις εργασίας, να βρούμε... Ε, ε, Παρακαλούμε, κυρία Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ για την ερώτηση, αλλά μάλλον θα έπρεπε να ρωτήσει η κυρία Μέρκελ και το λαό τη, γιατί πριν να λάβει αποφάσεις δεν είχε ρωτήσει αν ε, τη στηρίζει ο λαός της. Δεν μπορούμε τόσο ελευχαρά την καρδιά να χειριζόμαστε τέτοια προβλήματα. Κύριε Λάμπερτ, ένα λεπτό. Thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλοί σήμερα ανέφεραν τις λύσεις, όμως ξέρουμε ότι θα πάρουν καιρό οι λύσεις και εντωμεταξύ την κατάσταση του την πρέπει του πούσουμε άμεσα. Καλωσορίζω λοιπόν την αύξηση της χρηματοδότησης για το παγκόσμιο πρόγραμμα για τα τρόφιμα, αλλά πραγματικά σοκάρομαι. Σοκάρομαι που τόσα πολλά κράτη-μέλη πέρσι ε, περιέκοψαν και μείωσαν τη στήριξή τους για το παγκόσμιο πρόγραμμα για τα τρόφιμα, το επισητιστικό ε, πρόγραμμα. Βλέπουμε τόσοι άνθρωποι σε αυτή την, στον κόσμο να ζουν με μισό δολάριο την ημέρα. Τα κάτι μελη λοιπόν, ιδίω αυτοί που δεν πήραν μέρο στο πρόγραμμα αλληλεγγύη, θα έπρεπε να αισθανθούν όνειδο για το ε, πόνο που προκαλούν και την ταλαιπωρία. Σκεφτείτε πώς θα ζούσατε εσείς αν με τέτοιο ποσό έπρεπε να ζήσετε εσείς και οι οικογένειές σας. Άκουσα πολλούς να αναφέρουν και την Τουρκία ε, δεν είναι μια τρίτη χώρα ασφαλής για τους Κούρδους και θα πρέπει να στηρίζουμε τους Κούρδους και στην περιοχή του Εζαβάν και στην Τουρκία την ίδια, διότι είναι μέρος της λύσης. Και έπειτα θα πρέπει επιτέλου να υλοποιούμε τι αποφάσει που λαμβάνονται. Εάν θέλουμε να μιλάμε για του κανόνε και να πείθουμε ότι οι κανόνε αυτοί σωστώ προβλέπονται, θα πρέπει κάτι να κάνουμε και στην πράξη. Και να έχουμε και τι σωστέ πληροφορίε και τη σωστή ενημέρωση και τη διαδικασία ασύλου να αρχίζει τη στιγμή τη έλευση των προσφύγων. Όχι λίγε μέρε μετά όταν του έχουν ήδη ε, πιάσει η Frontex και ένα σωρό άλλοι οργανισμοί στα χέρια του. Ευχαριστούμε. Κυρία Λάμπερτ, υπάρχει ερώτηση για σας από την κυρία Γκραπίνη. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Γκραπίνη, την ερώτησή σα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφε, η κατάσταση είναι κατεπίγουσα και απαιτεί κατεπίγουσες λύσεις. Όντως, ε, είμαστε άνθρωποι και ανθρωπινά όντα όλοι μα. Ε, όμως δεν πιστεύετε ότι το Συμβούλιο θα έπρεπε να εξηγήσει σαφώ πώ αντιμετωπίσει τα γενεσιουργά αίτια αυτή τη κατάσταση, ώστε να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών για το πώ θα αποδεχτούμε του ανθρώπου αυτού. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο θέλουμε να μα πούνε πώ θα λύσουν και θα αντιμετωπίσουν τα αίτια όλων αυτών των προβλημάτων. Πρόεδρο, κυρία Λάμπερτ, την απάντηση. Ευχαριστώ. Σωστή ερώτηση. Νομίζω δεν ακούμε τα όσα πρέπει για το τι θα γίνει για την ειρήνευση τόπου και για τα άλλα αλληλένδετα ζητήματα που αφορούν ε, την δημοκρατία ή του πώς θα αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές στην περιοχή που αυτά όλα συμβάλλουν στην αστάθεια και ότι δεν κοιτάζουμε πραγματικά, όπως υπόθηκε προηγουμένως, πώς θα έχουμε μια συνεκτική πολιτική με κυβερνήσεις που καταπιέζουν τους ίδιους τους λαούς τους, τους ίδιους τους πολίτες τους, και στην ουσία βομβαρδίζουν τους πολίτες τους. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Μακ, για ένα λεπτό. Ε, όλοι συζητούν το ζήτημα της μετεγκατάστασης. Και όλοι θεωρούν ότι έχουν ηθικό πλεονέκτημα όταν κάνουν αυτή τη συζήτηση. Και δείχνουν με το δάχτυλο τις χώρες εκείνες που αρνούνται το σύστημα των ποσοστώσεων. Ενδιαφέρουσα ηθική, να προσπαθεί κανείς να είναι πιο ηθικός από τους άλλους. Αυτού του τύπου η αλληλεγγύη η οποία έρχεται επιβάλλεται δεν είναι στην πραγματικότητα αλληλεγγύη. Πρώτα ξεκινά η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστρέφει χώρες όπως η Συρία ή η Λιβύη. Μετά προσκαλεί τους πρόσφυγες στην Ευρώπη και μετά αξιοποιεί το σύστημα τους, ε, του Συμβουλίου για να αποφασίσει με ποιες ποσοστώσεις θα τους μετεγκαταστήσει. Ευελπιστώ ότι οι εκλογές στην Πολωνία θα δώσουν τη δυνατότητα να συνταχθεί αυτή η χώρα με την Τσεχία και τη Σλοβακία εναντίον αυτού του συστήματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ένα λεπτό, Άτκινσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Τούσκ αναφέρθηκε σε όλου του μετανάστε σαν να είναι πρόσφυγε. Δεν είναι όλοι. Κάποιοι ναι, κάποιοι όχι. Κάποιοι είναι οικονομικοί μετανάστε. Εκατοντάδε πρόσφυγε ε, στο Καλέ προσπαθούν να πεταβούν παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, και με την έλλειψη ελέγχου στα σύνορα φοβούμε για την ασφάλεια των Βρετανών πολιτών. Βάσει ε, τη Ευρώπη προσπαθούν, λένε Βρετανοί αριστεριστέ, να ε, δημιουργήσουν ε, αναταραχή στου καταβλισμού των προσφύγων και μας ζητάτε να αναλάβουμε και πάλι τον έλεγχο. Ενώ φαίνεται να ε, έχουν εγκληματική δράση οποιοδήποτε ε, πρόσφυγες ξεφεύγουν από τους καταπλησμούς, δημιουργούν προβλήματα στα τούνελ ε, και αναταραχές. Ουγγαρία με τον κύριο Ορμπάν δείχνει ότι ε, μπορεί να λάβει μέτρα και να είναι ένας καλός Ευρωπαίος που ε, κάνει ό,τι θέλει ε, ερχόμενος εδώ να απευθυνθεί στο Κοινοβούλιο και επιβάλλοντας τη δική του ατζέντα. Ε, Όμως ε, δεν είναι έτσι και δεν μπορούμε να καλούμε του υπόλοιπου Ευρωπαίους να, συμπεριφερθούν, να συμπεριφερθούν ανάλογα. Θα πρέπει κύριε Πρόεδρε να ξαναχτίσουμε τα τείχη στην Ευρώπη λοιπόν και να ισχύει απολύτω το Δουβλίνο. Κύριε Λαμασούρη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε γίνεται μία επίδειξη εδώ. Αφήστε τα κρατημέλη ακόμα και τα πιο ε, δυνατά αυτά που θέλησαν να μείνουν εκτό του Σέγγεν να λύσουν μόνοι του το πρόβλημα των μεταναστών δεν γίνεται. Οι, πανικό, οι λύσεις του πανικού φαίνεται να αγγίζουν το γελίο, το καταγέλαστο και κάποιες φορές και το ε, αποτρόπαιο. Εδώ βλέπουμε ότι τα μέτρα που έχουμε λάβει δεν είναι σωστά. Η μαζική έξοδος των πολιτών προς την Ευρώπη έχει να κάνει με τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία. Και μόνο αν τεραμετιστεί αυτός θα τερματιστεί και η έξοδος. Βλέπουμε ε, εκατοντάδες χιλιάδες νέοι, πολλές φορές ολόκληρες οικογένειες από την Αφρική και την Ασία, ε, τα μέσα στη Μέση Ανατολή, να προσπαθούν να σωθούν φτάνοντας στην Ευρώπη μέσω των Βαλκανίων ή τη Σικελία πριν από τις Κανάριες νήσους. Αυτό δεν θα πάψει μεταναστευτικέ οδοί θα είναι μια σταθερά των ε, αιώνων αυτών. Και αυτοί που ρίχνονται στο δρόμο είναι όσοι δεν βρίσκουν ότι έχουν μέλλον στο σπίτι τους. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει σωστή κατανομή των ετών ασύλου και να μην είναι κάτι που θα το, θα, το θα το αποφασίσουμε μόνο σε καταστάσεις ε, όπου φτάνουμε να υποφέρουμε. Θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερή διαρκής πολιτική για το άσυλο και τους μετανάστες, μια εξωτερική πολιτική κατάλληλη ε, γιατί την έχει ανάγκη όλη η Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δίκιο να ε, θέτει τα θεμέλια και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έπρεπε μεγάλο σφάλμα εάν δεν έφερνε εις πέρας αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Γκυγιόμ για 1,5 λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Όλοι συμφωνούν ότι το Συμβούλιο της 23ης Σεπτεμβρίου, όπως και το ΤΣΑΙ της 22ης επέτρεψε έστω και επώδυνα να προχωρήσουμε σε κάποια σημαντικά βήματα ω Ένωση για την αντιμετώπιση τη κρίση των προσφύγων, αλλά πρέπει αυτό να εγγραφεί μέσα σε, ένα, σε μια πολύ πιο περίπλοκη και πιο πλήρη διαδικασία και διαδρομή. Δεν πρέπει να λησμονήσουμε το ουσιώδε. δηλαδή πρέπει να δράσουμε κατεπηγόντω γιατί το απαιτεί η ανθρωπιστική κατάσταση, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δώσουμε προοπτικέ και μέσα για, τη μακροπρό... για το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και την αντιμετώπιση του κλίματος. Ω εκ τούτου έχω τα εξή ερωτήματα προ την Επιτροπή και το Συμβούλιο. τα λοιπόν όλο και πιο κατεπίγουσα για αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και τις κινήσεις. Θέλουμε να έχουμε περισσότερη κοινοτικοποίηση, δηλαδή των αποφάσεων και των πρακτικών μας. Δεύτερον, τα λειτουργικά ζητήματα απαιτούν και τη χρηματοδότηση, βράχη, μέσο και μακροπρόθεσμα. Εδώ το θέμα του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Θεωρείτε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να πτήσουμε μια πολιτική ευρωπαϊκή με τον υφιστάμενο ευρωπαϊκό προπολογισμό. Και τρίτον, η εξωτερική διάσταση, αυτό που λέγεται δηλαδή για την περίπτωση τη παροχή του διεθνού προστασία σε κάποιου, σε εξωτερικέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί θα του σταθεροποιούμε του πρόσφυγε. Αυτό πώ θα γίνει, με κάποια αιγίδα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Κυρία Γκυλιόμ, έχετε μπλε κάρτα. Βίμπεργκερ, έχετε το λόγο για την ερώτηση προς την κυρία Γκυλιόμ. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γκυλιόμ, λέτε να γίνεται υποχρεωτική κατανομή των προσφύγων αυτών, αλλά κλείσει το θέμα των 160.000 προσφύγων και τους κατανείμουμε, θα έρθουν και άλλα προβλήματα. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους τι θα τους κάνουμε μετά, τους 500.000 που θα έρθουν και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Απάντηση. Κυρία Βίνμπεργκερ, ε, είχαμε πολλέ συνεδριάσει υπό Επιτροπή των Πολιτικών, της Επιτροπής των Πολιτικών Ελευθεριών και εκ μέρου και τη ομάδα μου. Ποτέ δεν δέχθηκα να υποβιβάσω το πρόβλημα. Δηλαδή, πρέπει να δώσουμε απάντηση στην ανθρωπιστική κρίση, όπω είπα, αλλά πρέπει να δώσουμε και αποφάσει μακροπρόθεσμε για την αντιμετώπιση του προβλήματο. Δηλαδή, πρέπει να κοιτάξουμε την πηγή των τερνόμενων προβλημάτων ε, σε σχέση με τα κράτη από τα οποία προέρχονται οι πρόσφυγε. Και βεβαίω υπάρχει και το ζήτημα τη ενσωμάτωση και, κυρία συνάδελφε, διαφωνούμε διαφωνούμε απολύτω ω προ τι πολιτικέ ενσωμάτωση που προβλέπετε, γιατί εσεί δεν προβλέπετε ουδέμια πολιτική ενσωμάτωση. Ευχαριστώ, Σούλικ. Ένα λεπτό. Το καλοκαίρι γινόταν λόγος για 800.000 πρόσφυγες που θα έφταναν φέτος στη Γερμανία. Τώρα έχουμε φτάσει του υπολογισμούς στο 1,5 εκατομμύριο. Η απόκληση αυτή, 700.000 πρόσφυγες, πρέπει να χρεωθεί στην Άγγελα Μέρ και την ανεύθυνη καταστροφική πολιτική της. Η κυρία Μέρκελ έθεσε εκτός λειτουργίας, εκτός ισχύω το σύμφωνο του Δουβλίνου. Δεν μπορεί να πράττει κάτι τέτοιο. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους αυτούς είναι οικονομικοί μετανάστες και όχι πρόσφυγες λόγω πολέμου. Εάν λοιπόν μπορεί κανείς να περάσει από τόσες ε, περιπέτειες για να φτάσει κάπου, προσφανώς δεν είναι πρόσφυγες. Και ξέρουμε ότι αυτοί οι πρόσφυγες θα κάτσουν στη Γερμανία να δουλέψουν για να πληρώνουν τις συντάξεις των Γερμανών συνταξιούχων. Είναι μεγάλος ο φραγμός ε, του ελάχιστου μισθού και η Γερμανία μπορεί να προσφέρει κοινωνικές ε, παροχές. Η κυρία Μέρκελ όμως λησμονεί ποιος την έχει εκλέξει και ποιον οφείλει να προστατέψει. Τώρα έχει έρθει η ώρα να σταματήσει αυτή η ε, εισβολή, όπως έπραξε η Αυστραλία. Ευχαριστώ. Εύα Ζολή, ένα λεπτό έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως θα την ήθελα, όπως όλοι θα τη θέλαμε, να επιδεικνύει αλληλεγγύη, αυτή η Ευρώπη δεν υπάρχει. Αυτό είναι το συμπέρασμα από αυτό το τραγικό σε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23 η Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπερψηφίσει έναν προσωρινό μηχανισμό ε, μετεγκατάστασης όπως τον έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε συνολικά όλα τα κράτη-μέλη με αξιοπρέπεια και με αλληλεγγύη να ανταποκριθούν σε αυτή την προσφυγική κρίση. Ανταυτού τα κράτη-μέλη ε, αποδεικνύονται έτσι, να, ότι υπολογίζουν και προσπαθούν να βρουν ποιο να επιωφεληθούν από αυτή την κρίση. Χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση με πολιτική βούληση και με θάρρος. Μετά την κρίση στην Ελλάδα, της Ελλάδας, η κρίση των προσφύγων, η προσφυγική μας αποδεικνύει τις ελλείψεις της Ευρώπης. Δεν έχουν άλλη υπομονή οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πηγαίνουν προς τα άκρα. Γιατί αυτή η ελπίδα την οποία περίμεναν από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, αποδεικνύεται στην πράξη. Ας ξυπνήσουμε. Κυρία Ζολή, υπάρχει μια ερώτηση προς εσάς από τον κύριο Κάρβερ. Ευχαριστώ κυρία Ζολή. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν, ε, όπως θα τη θέλατε δεν υπάρχει. Αλλά ακριβώς αυτό δεν είναι το πρόβλημα ότι πρόκειται για μια οτοπία αυτό που θα θέλατε. υπάρχουν τα κράτη-μέλη. Και ακόμα και αν δεν σας αρέσει αυτό, τα κράτη-μέλη υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους. Και αυτό πάντοτε έτσι θα είναι. Επομένως, τι περιμένετε να γίνει, πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί στην πράξη του σχέδιό σας μέσα στην πραγματικότητα. Κυρία Ζολή. Η κρίση η προσφυγική είναι αποτέλεσμα του χάους που υπάρχει στον κόσμο. Που είναι αποτέλεσμα Τη εξωτερικής μα πολιτικής ή μάλλον της απουσίας εξωτερικής πολιτικής από την πλευρά τη Ένωση. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε μια έκτακτη ανάγκη την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, όπως το είπε και η συνάδελφός μου. Ανταυτού βλέπουμε τα κράτη-μέλη να μειώνουν τη συμμετοχή τους στα ανθρωπιστικά ταμεία, στο παγκόσμιο επιστημιστικό πρόγραμμα, το οποίο δεν έχει πλέον τους πόρους που χρειάζεται για να παρέχει την επιστημιστική βοήθεια που χρειάζονται οι άνθρωποι αυτοί. Κύριος Μάγερ, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, οι Βρυξέλλες με δικτατορικό τρόπο αποφάσισαν να μετατραπεί η Ευρώπη σε ένα μεγάλο καταβλισμό προσφύγων. Η κατανομή 160.000 προσφύγων ανήκει το νασκό του αιώλου. Δεν έχουμε καν δει τι συνέπειες έχει αυτό. Τώρα αρχίζει το πανηγύρι. 600.000 έχουν φτάσει με τα πρόσφυγες παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έρθουν και πολλοί άλλοι ακόμα. Πρέπει λοιπόν ε, να βρούμε μια, έναν τρόπο πραγματικής δημοκρατικής και ευρωπαϊκής άμυνας για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Το 60% των ε, Ολλανδών θεωρούν ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε τόσους πρόσφυγες. Πολλοί είναι και οι Γερμανοί και η πλειονοψηφία τους μάλιστα, όπως και οι Αυστριακοί που θεωρούν ότι δεν ε, πάει άλλο. Κύριε Πρόεδρε, φτάνει πια δεν μπορούμε να δεχθούμε ούτε έναν παραπάνω πρόσφατα. Πρέπει να κλείσουμε τα σύνορά μα. Ο μόνο τρόπο είναι αυτό. Ονορεύολε Μάιερ. Κυρία Μάιερ, έχετε μπλε κάρτα από τον κύριο Ούρμπαν Κρέστο, αν τη δέχεστε παρακαλώ. Με εντυπωσιάζει η ελαφρότητα με την οποία μιλάτε εδώ μέσα για κατάρες για τσουνάμι, για εισβολές. Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, γιατί τροφοδοτείται με τα λόγια αυτά τον ε, ρατσισμό και την ξενοφοβία εις βάρος των ανθρώπων αυτών προσπαθούν να ξεφύγουν από τις βόμβες, από το θάνατο, από την εξαθλίωση. Όταν, σας, όταν καλείτε άλλους να επιβάλλουν ε, πολιτικές λιτότητας, δεν σας είδα να φωνάσετε τόσο δυνατά. Στα ανθρώπινα δικαιώματα όμως μιλάτε για πλήγια στο φαράω. Δεν καταλαβαίνετε ότι καταστρέφετε την Ευρώπη των αξιών και χτίζετε την Ευρώπη της ξενοφοβίας. Παρακαλώ κύριε Μάιγερ. Ναι, σας επιστρέφω τα, ή μάλλον τα αγνοώ τα σχόλια περί ρατσισμού και ξενοφοβίας. Δεν έχετε ιδέα για το τι συμβαίνει στις κάτω χώρες. Δεν είμαστε κοντά στην Τουρκία και τη Μεσόγειο. Αυτό που αναζητούμε λοιπόν είναι να εξασφαλίσουμε να ε, κρατήσουμε την ασφάλεια για τους Ολλανδούς γιατί ξέρετε αυτοί οι άνθρωποι έρχονται να βρούνε όχι ασφάλεια από τον κίνδυνο του πολέμου αλλά δωρεάν επιδοτήσεις, δωρεάν επιδόματα και στέγη. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι που δεν θέλουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κεφαλό Γιάννη, 1 και 30 παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποδέχτης τεράστιου αριθμού μεταναστών και προσφύγων. Η διπλή αυτή κρίση είναι πρόβλημα ευρωπαϊκό και χρειάζεται ευρωπαϊκή προσέγγιση, αλληλεγγύη και υπευθυνότητα. Είναι επομένω επιτακτική ανάγκη στήριξη στα κράτη-μέλη πρώτη γραμμή όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα. Είναι επιτακτική ανάγκη της παροχής τεχνικής και οικονομικής βοήθειας στις χώρες εισόδου, παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε μετανάστες και πρόσφυγες. Ο Φούρναρης από την κόνηση της Ανατολικής Ευρώπης είχε αναφερθεί ο πρόεδρος Γιούγκερ στην περίπτωσή του είναι χαρακτηριστική των αρχών και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των λαών της Ευρώπης η λύση δεν είναι εύκολη. η ευρώπη πρέπει να δράσει προληπτικά να στρέψει την προσοχή της στις χώρες διέλευσης όπως παραδείγματος χάρη η τουρκία να στρέψει την προσοχή της στις χώρες προέλευσης των μεταναστών και βεβαίως σε επιχειρησιακό επίπεδο χρειάζεται καλύτερη επιτήρηση των συνόρων εντοπισμός των παράνομων κυκλωμάτων των μεταναστών και η ενίσχυση της frontex η ευρωπαϊκή ένωση και θέλει και μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία αυτή τη μεγάλη πρόκληση. έχουμε εμπιστοσύνη σε εσά κύριε juncker και κύριε tusk πιστεύουμε ότι η ευρώπη και σε αυτή τη μεγάλη κρίση θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει με βάση την ιστορία και τις αρχές. σας ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ε, ε, ευχαριστώ. Κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε μία ερώτηση από τον κύριο η ερώτησή σας, παρακαλώ. E, Ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Λαμασούρ, αλλά ευκαιρία είναι να ρωτήσω με συγχωρείτε, συγχωρείτε. Είχαμε καταλάβει από την γραμματεία ότι θέλατε να κάνετε ερώτηση προς τον κύριο Κεφαλογιάννη. Δυστυχώς δεν γίνεται να θέσετε ερώτηση έτσι γενικώ. Για γαλάζια κάρτα μιλούσαμε. Όχι, όχι, δεν γίνεται έτσι. Κυρία Τόγια, κυρία Τόγια για 1,5 λεπτό. Ε, με το Συμβούλιο του Σεπτέμβρη ξεκίνησε η πραγματική δουλειά πρέπει πολύ γρήγορα να αντιμετωπίσουμε τα εξή θέματα. Hot spot, έλεγχο, γρήγορη εξέταση των ετοιμάτων, επανεγκατάσταση και επαναπατρισμό όποτε χρειαστεί. Όλα αυτά να λειτουργήσουν ταυτόχρονα γιατί είναι αλληλένδετα. Χρειάζεται λοιπόν η ευρωπαϊκή δράση να είναι αποτελεσματική και να σέβεται τα δικαιώματα και την, ε, τον ανθρώπινο πόνο αυτών των ε, προσφυγών. Κύριε και μια ερώτηση προ εσά. Ευχαριστώ για την αποφασιστικότητα και την πυγμή με την οποία δράσατε. Να συνεχίσετε, σα παρακαλώ. Στον ε, πρόεδρο Τούσκ να απευθύνω το εξή κάθε σεβασμό, μιλάτε για τι ε, τεράστιε ευθύνε σα, αλλά χρειαζόμαστε μια δράση πιο αποτελεσματική και έναν ρόλο σα πιο αποφασιστικό για να πείσετε το Συμβούλιο, εφόσον εσεί οδηγείτε και πρέπει να αναλάβουν τι ευθύνε και την ελληνική που αναφέρατε και στην παρέμβασή σα. Εσεί πρέπει να κάνετε αυτά τα βήματα ε, που πρέπει να συμπαρασύρουν το Συμβούλιο. Στην ομιλία σα ε, κατανείματε κάποιε ευθύνε και βάλατε στο ίδιο επίπεδο χώρε όπω η Ιταλία και η Ελλάδα με χώρε που δεν θέλω να αναφέρω αλλά που σηκώνουν τους ώμους και εδώ και τρία με πέντε χρόνια κάνουν ε, μαθήματα ή βάζουν στη φυλακή όποιον βρίσκουν ε, ανυπεράσπιστο και δεν δίνουν ένα καλό παράδειγμα για το καλό όνομα της Ευρώπης. Πώς μιλάτε λοιπόν για τις ευθύνε της Ιταλίας. Εμείς μεταξύ της ευθύνη και της ζωής ε, αποφασίσαμε να διασώζουμε παιδιά, γυναίκες και άντρες όπως θα έπρεπε να κάνετε και εσείς. Ευχαριστούμε κυρία Τόγια. Διέλη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε για να δώσει τέρμα σε αιώνες πολέμων στους εθνικούς εγωισμούς και τον στήρο ανταγωνισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών εθνών. Υποτίθεται ότι έχει χθιστεί σε βάση κοινών αξιών αλληλεγγύη και αλληλοσυνεργασία. Θα πρέπει λοιπόν μια Ευρώπη 500 εκατομμυρίων πολιτών να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή τη μεταναστευτική κρίση. Εάν υπάρχει τέτοια ένωση βεβαίως. Αλλά εδώ μιλάμε για μια Ευρώπη που ασθενεί και εφόσον υπάρχει νόσος θα πρέπει να σκεφτούμε ποιοι είναι οι ιοί που την απειλούν. Υπάρχει ένας ιός που έχει μολύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ιός αυτός είναι η εγωπάθεια των πολιτικών ηθινόντων προσπαθούν να παίξουν τα δικά τους πολιτικά παιχνίδια εσωτερικώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Γιούνκερ, συμφωνήσαμε για δύο πράγματα ήδη πριν το καλοκαίρι και μας υποσχεθήκατε μέτρα ε, ήδη το Σεπτέμβριο. Πού είναι αυτά τα μέτρα. Η Ουγγαρία δεν είναι μόνο ο κύριος Ορμπάν και η κυβέρνησή του, είναι και άλλοι άνθρωποι. Ε, είναι και δεκάδες ε, χιλιάδες πολίτε και εθελοντέ που βοήθησαν του πρόσφυγε και πολλοί είναι εδώ στην Ολομέλεια ω προκεκλημένοι. Αυτή είναι το μέλλον τη Ευρώπη. Σα ευχαριστούμε. Η... Κύριε Βιέλη, υπάρχει ερώτημα για σας. Από την κυρία Μορδάη, παρακαλώ, η ερώτησή σας. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με, το, με την ερμηνεία, θα το λύσουμε αμέσως. Πρόεδρε, Εσεί που είσαστε υπεύθυνοι να λαμβάνετε τι αποφάσεις για το θέμα τη μετανάστευση. καλό θα είναι να αντιληφθείτε ότι όλοι αυτοί που ζουν στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολα σχέση με τη μετανάστευση και την έλευση των μεταναστών. Καλό θα ήταν ε, να προσφέρετε με τις γνώσεις σας ε, ε, λύσεις και να βοηθήσετε στην εξέβριση σωστών λύσεων. Ευχαριστώ. Ήμουν μέλος του Γκρικού Κοινοβουλίου και όντως την κρίση των μεταναστών Μιλάμε για ένα hot spot, κάποιες εκατοντάδες χιλιάμετρα από εκεί που ο κύριος Ορμπάν ε, άρχισε να χτίζει αυτό το τείχος μαζί με τους δικούς του συνεργάτες. Κυρία Μορβάη, ξέρετε ότι η κοινωνία των πολιτών, οι άνθρωποι, οι απλοί θα μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα με τρόπο απλούστερο αν δεν υπήρχε αυτή η πολιτική εκστρατεία από τον κύριο Ορμπάν και εσείς είστε από κόμμα της ακροδεξιάς, θύντες ε, και ε, οι δυνάμεις της. Αυτό είναι το κόμμα που έχουν αμαυρώσει την εικόνα της Ουγγαρίας. Επιστρέψτε πια στην ε, λογική της ελληνικής. Ευχαριστούμε κυρία Γκόμες για ένα λεπτό. Όχι κύριε Τούσκ, το οχυρό της Ευρώπης που θέλετε να δημιουργήσετε δεν θα προστατεύσει τους, Ευρω... τους Ευρωπαίους. Ε, το, οι κυβερνήσεις και το Συμβούλιο εδώ και πολύ καιρό δεν έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια πολιτική για να αντιμετωπίσουν τη ροή των μεταναστών. Δεν ανοίγουν νόμιμες οδούς ασφαλείς για να μην συνεχίσουμε να τροφοδοτούμε την εμπορία ανθρώπων και τους διακινητές και δεν έχουμε μια πολιτική, διπλωματική και στρατιωτική σωστή για να αντιμετωπίσουμε τα αίτια της κρίσης, τον πόλεμο στη Συρία, ε, τα όσα συμβαίνουν στη Λιβύη και την επέκταση του Ισλαμικού κράτους. Εδώ βλέπουμε λοιπόν κονδύλια να δαπανώνται στην πολιτική γειτονία, ε, αντί να δημιουργούμε σχολεία για τα παιδιά και τους νέους ε, στους καταπλησμούς των προσφύγων. Τα ευρωπαϊκά κράτη αντιδρούν με τρόπο εθνικιστικό. Αμαυρώνουν την εικόνα της Ένωσης αντί να έχουν μια ε, ε, συντονισμένη εξωτερική και εσωτερική πολιτική. Ε, έτσι εξυπηρετούμε τους τρομοκρατές οι οποίοι θέλουν να υπονομεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουν μόνο επιλύονται με στρατηγική σύγκληση, με κατανομή και συνεργασία, με εξωτερική πολιτική ασφάλειας και άμυνας που είναι κοινέ. Δεν μπορούμε διαρκώς να ζητούμε εξαιρέσεις από το Συμβούλιο. Χρειαζόμαστε περισσότερη ένωση και όχι περισσότερα τύχη. Ευχαριστούμε κυρία Γκόμες. Ε, μία ερώτηση προς εσάς. Τη δέχεστε από τον κύριο Βάγκλ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συνάδελφε, συχνά ερχόμαστε αντιμέτωποι με προβλήματα διεθνών διαστάσεων. Υπάρχουν πολλές ε, τάσεις κερδοσκοπίας ε, και υπάρχουν και πολλέ εικασίε για το τι ε, διαφεύγουν αυτοί οι άνθρωποι από τι χώρε του. Οι περισσότεροι διαφεύγουν από συνδικέ πολέμου. Ισχύει αυτό σαφώ για την Συρία. Πρέπει όμω να καταλάβουμε ότι και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει ανανεωμένε υποχρεώσει για να διατηρεί την ειρήνη. Θα πρέπει να είναι αποτελεσματικότερη στην επαναγκατάσταση ε, ε, των ανθρώπων αυτών και θα πρέπει να είναι αποτελεσματικότερη στην ειρηνική επίλυση των προβλημάτων. Πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία στην ειρήνη. Παρακαλώ, κυρία Γκόμος. Κόμες. ευχαριστώ. Ε, αγαπητέ συνάδελφοι, έχετε δίκιο. Ακριβώ γι' αυτό ζητώ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο οι κυβερνήσει να πάψουν. Να πάψουν να μποϊκοτάρουν το κοινό πλαίσιο για την κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα και την κοινή πολιτική άμυνα. Τι χρειαζόμαστε και πρέπει να έχουμε στατική δράση. Μόνο συντονισμένοι μπορούμε να αλλάξουμε κάτι, να πάψουμε τον πόλεμο στη Συρία και όχι να επιδεινώνουμε τα πράγματα όπω θα γινόταν με μια νίκη του Ασάντ. Και εδώ θα πρέπει να σταματήσουμε μπορέσουμε να πάψουμε να ε, υπονομεύουμε ε, όσους ε, προσπαθούν να αγωνιστούν κατά του Ισλαμικού κράτους στο βόρειο Ιράκ, να και την Πεσμέρκα και να έχουμε μια συντονισμένη δράση και εδώ. Δεν μπορούμε να απογοητεύουμε διαρκώ του πολίτε. Δεν μπορούμε να υπονομεύουμε την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών μα χωρί να αντιμετωπίζουμε τα γενεσιουργά αίτια των όσων αναγκάζουν του ανθρώπου να δραπετεύουν, να ε, γλιτώνουν από τη Συρία, την Ερυθρέα και αλλού. Ευχαριστώ. Να θυμίσω στους συναδέλφους ότι στο τέλος της πρωινής συνεδρίασης έχουμε και τις ψηφοφορίες μετά από αυτή τη συζήτηση. Και έχουμε και άλλη συζήτηση μετά από αυτήν. Θα παρακαλέσω λοιπόν να σέβεστε λίγο τα χρονικά όρια. Ο κύριος Μαυρίδης για ένα λεπτό παρακαλώ. Το ανθρωπιστικό πρόβλημα κύριε Πρόεδρε είναι η είναι η διάσωση των ανθρωπίνων ζώων. Αλλά μπορεί κάποιος να διανοηθεί ασφάλεια και προστασία για αυτούς τους φιλήσυχους πληθυσμούς ενώ όσο δεν υπάρχει εκρίζωση πρώτα απ' όλα του ISIS και αυτό απευθύνεται και στον κύριο Τούσκ ειδικά προσωπικά για τα σχόλια που έκανε προηγουμένως η ευρωπαϊκή μας συνείδηση μας επιβάλλει να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες αλλά πρέπει να βοηθήσουμε να σταματήσουν να υπάρχουν πρόσφυγες και αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς εκρίζωση του isis. απεχθάνουμε τον ασαντ αλλά έχουμε προτεραιότητες. ο ερντογάν που επισκέφτεται τώρα τις βρυξέλλες καταδιώκει τον τύπο τους πολιτικούς του αντιπάλους βομβαρδίζει τον κουρδικό πληθυσμό συνεχίζει την παράνομη κατοχή ευρωπαϊκών αλλά κρίνουμε εδώ ότι για υπέρτερους λόγους τον έχουμε ανάγκη. μιας και βρίσκεται στις βρυξέλλες αντί τις συναλλαγές που κάνουμε μαζί του τουλάχιστον ζητήστε του να σταματήσει να βομβαρδίζει τους κούρδους. μια τελευταία φράση αυτό που μας διαφοροποιεί εμάς στην Ευρώπη είναι τα συμφέροντά μας, είναι και οι αξίες μας. Onorevole Tonino Pizzua, per un minuto. Prego. Hola, Presidente. Gospodine Juncker. Ευχαριστούμε, κύριο Τονίνο Πιτσούα, για το Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 29 κράτη-μέλη. Όμως η επικράτη αυτή δεν είναι φανταστική. Βλέπουμε πόσοι είναι οι πολίτε που είναι άνεργοι ε, και δυστυχεί σε αυτή την Ήπειρο και βλέπουμε ότι φτάνουν στι ίδιε καταστάσεις, ε, στις ίδιε συνθήκε ζωή με του ε, πρόσφυγε Εδώ μιλάμε για μια διεθνή κρίση, όχι μόνο για μια κρίση προσφύγων. Αυτό φαίνεται από τα όσα συμβαίνουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαίνεται να μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Ιταλία, ε, λόγου χάρη και Γερμανία, δέχονται το μεγαλύτερο ποσοστό, τη μερίδα του λέοντος των προσφύγων. Αυτό δείχνει ότι μπορούμε να λειτουργούμε καλά ως Ευρωπαϊκή Ένωση υπό κανονικές συνθήκες, αλλά όχι σε έκτακτες. Η Κροατία είναι ένα από τα κράτη που έχουν εκτεθεί στην κρίση των προσφύγων, αλλά δεν είναι μέλος του χώρου του Σέγγεν. Χρειάζεται λοιπόν το αλληλεγγύη, διότι αντιμετωπίζουμε πολιτικούς εκπομπισμούς, στατιτικοποίηση των συνόρων μας ε, και ε, τάσεις ε, ακραίες σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να δούμε τι είδους κοινωνίας θέλουμε να δημιουργήσουμε για να ζούμε σε αυτή και τι είδους εικόνα θέλουμε να δείχνουμε στον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστούμε. Υπάρχει ερώτηση για τον κύριο Πιτσούα. Όχι, ωραία. Ο κύριος Ιγκλέσιος για δύο λεπτά. Θα μιλήσατε προηγουμένω, αλλά τώρα παίρνετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αλλά ανακατεύομαι να σας ακούω να μιλάτε ορισμένοι εδώ στην αίθουσα για πληγή, για ασφάλεια και όλα αυτά. Είναι προσβολή για τη δημοκρατία και για το σώμα. Όταν μιλούμε για ευρωπαϊκές αξίες, ένα πράγμα μόνο μπορούμε να σας χαρακτηρίσουμε. Είστε σκουπίδια, σκουπίδια που μιλάτε έτσι για ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από την εξαθλίωση και από τον πόλεμο. Η απάντηση λοιπόν σε όλα αυτά που λένε τα σκουπίδια είναι μία. Τα τελευταία 15 χρόνια η ευρωπαϊκή πολιτική δεν συνέβαλε παρά μόνο στο να ρίχνει λάδι στη φωτιά. Κανείς δεν λέει εδώ ότι το πρωτόκολλο του Δουβλίνου επί παραδείγματι θα επέτρεπε με την κατάργησή του μόνο να αποτραπούν τέτοιου είδους εικόνες, να μην βλέπουμε παιδιά νεκρά πάνω στις παραλίες. Απέναντι λοιπόν στα σκουπίδια ας είμαστε λιγότερο υποκριτές. Κύριε Ιγκλέσιας, έχετε μια μπλε κάρτα. Κύριε Ιγκλέσιας, δέχεστε την ε, ερώτηση. Le Breton. Τη δέχεστε. Ευχαριστώ που δέχεστε την ερώτησή μου. Αγαπητέ συνάδελφε, με ξαφνιάζει το γεγονός ότι χαρακτηρίζετε σκουπίδια ορισμένους από τους συναδέλφους σας εδώ στην Ολομέλεια. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και δεν νομίζω ότι μπορούμε να το εξαντλήσουμε στην ανταλλαγή Ιβρεών. Δεν δέχεστε ότι είναι μαζική αυτή η μετανάστευση, ότι ο όγκο τη ξεπερνάει αδίποτε προσδοκία και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να μιλούμε για ρατσισμό και ξενοφοβία. Πρέπει να ανησυχούμε κιόλα. Γι' αυτό λοιπόν πέραν των Ιβρεών σα. δεν θεωρείτε ότι τα κράτη έχουν κάποιο δίκαιο που ανησυχούν για τα συμβαίνοντα. Δεν ε, θεωρείται ότι πρέπει να προσπαθήσουν να περιορίσουν τις ροές των προσφύγων τα κράτη και δεν θεωρείται, ζητώ τη γνώμη σας, ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να σταθεροποιηθούν αυτές οι ροές των προσφύγων στις χώρες όπου βρίσκονται και να μην φτάνονται μέχρι εδώ. Να μην ανοίγουμε δηλαδή τις πόρτες όπως έκανε η κυρία Μέρκελ με τις δηλώσεις της. Κύριε Ιγλέσιας, έχετε το λόγο. Είστε Ευρωπαίος κύριε συνάδελφε και θέλετε να μάθετε μήπως ε, πως ε, οι παππούδες σας όπως και οι δικοί μου άλλωστε αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους. Εγώ αποκαλώ σκουπίδι ή ονδήποτε επικαλείται τη μνήμη των παππούδων μας για να μιλήσει για πληγή για να μιλήσει για κατάρα και για εισβολή. Δεν μπορούμε λοιπόν με τον εγωισμό να απαντάμε σε ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να ξεφύγουν από την καταστροφή. Δεν είναι αυτή η δημοκρατική Ευρώπη που προσπαθούμε να χτίσουμε. Τώρα θα ακούσουμε τις απαντήσεις των πρόεδρων Ιούνκερ και Τούσκ, αλλά πριν ξεκινάει η διαδικασία Catch the Eye. Βλέπετε το χαρτί, έχουν στήσει πάρα πολλοί συνάδελφοι το λόγο. Δεν θα μπορέσω να δώσω το λόγο παρά μόνο σε έναν συνάδελφο αναομάδα δεδομένου και του χρονικού περιθωρίου που έχουμε. Ξεκινά ο κύριος Μπόγκοβιτς για ένα λεπτό και παρακαλώ να τηρούνται οι χρόνοι. Κύριοι συνάδελφοι, η Ευρώπη δεν θα αναλάβει στους ώμους της το σύνολο του προσφυγικού προβλήματος του κόσμου γιατί ε, δεν το προκάλεσε. Είμαστε ε, μέρος της λύσης αλλά όχι εμείς ο μεγάλος ασθενής. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ένωσης και αυτές πρέπει να γίνουν σεβαστές. Και αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα συζητούμε και στο εσωτερικό των χωρών μας. Σε διάφορα κράτη του κόσμου έπεσαν τα καθεστώστατα και αντικαταστάθηκαν από γεωδικτάτορε που δεν έχουν κανένα σεβασμό για την ανθρώπινη ζωή και έτσι προέκυψαν όλοι αυτοί οι πρόσφυγε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε πάνω απ' όλα. Πρέπει να προσφέρουμε βοήθεια σε αυτέ τι χώρε και μόνο ε, ε, με την ειρήνη μπορεί να επιληθεί τελικά το πρόβλημα. Γνωρίζουμε ότι η μεταναστευτική κρίση θα συνεχίσει εξαιτίας της δημοκρατικής αύξησης ε, στην ε, Αφρική, για παράδειγμα. Το οποίο σημαίνει ότι όσον αφορά τους μετανάστες χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμες λύσεις. Πρώτα απ' όλα ξεκινώντας, βοηθώντας αυτούς που βρίσκονται ήδη στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ε, από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτες που το λόγο κύριο Τζουφρίντα. Η κυρία Τζουφρίντα, παρακαλώ. Αμέσω μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στι 23 Σεπτεμβρίου, που ε, ήταν ε, πολύ πιο δύσκολη ακριβώ επειδή την αναβάλαν για καιρό, νομίζω ότι πώ θα μπορέσουμε όλοι μα από κοινού να πούμε ότι πρέπει οι Ευρωπαίοι πολίτε να συνεχίσουν να πιστεύουν στι ευρωπαϊκέ αξίε, εάν δεν είχαμε φτάσει έστω σε αυτό το αποτέλεσμα εδώ, στο Ευρωκοινοβούλιο, με μεγάλη πλειοψηφία επανειλημμένω ε, Είμαστε υπέρ του βήματος αυτού που είναι μόνο ένα πρώτο βήμα παρά την αποφασιστικότητα και την που επιδείχθηκε. Εδώ χρειάζεται μια διαδικασία με συγκεκριμένες χειροπιαστές πράξεις που να λαμβάνουν υπόψη τις σοβαρότατες γεωπολιτικές αλλαγές που προκαλούν τις μεταναστευτικές, ροές και που δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με τον τρόπο του παρελθόντος. Εδώ χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα, διαδικασία ένταξης των προσφύγων, κάτι που θα πρέπει να μας κάνει να προβληματιστούμε εντός της Ευρωπαϊκής παρά την αντίθεση και την ε, δρυμή αντιπαράθεση κάποιων χωρών. Αυτές θα πρέπει να μας οδηγήσουν να συλλογιστούμε και να κάνουμε τα ανάλογα βήματα. Οι δηλώσεις του Πρόεδρου Γιούνκερ για την κατάσταση στην Ένωση υπογραμμίζουν ότι δεν είναι αυτό αυτό που λείπει μάλλον πάνω απ' όλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ένωση. Ο κ. Μαριά, για ένα λεπτό. Χιλιάδε πρόσφυγε κατακλείζουν την Νότια Ευρώπη και κυρίω την Ελλάδα που δεν αντέχει άλλους πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες. μέχρι σήμερα έχουν εισέλθει στην πατρίδα μας πάνω από 260.000 πρόσφυγες. ο κόμπος λοιπόν έχει φτάσει στο χτένι και πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα. πρώτον ανάληψη πρωτοβουλειών για την εμπέδωση της ειρήνης στη μέση ανατολή και τη βόρεια αφρική να διαμενηθεί στην τουρκία ότι πρέπει να σταματήσει να εμπορεύεται την αγωνία των προσφύγων και να σταματήσει να υποθάλπει τα δουλεμπορικά κυκλώματα να καταργηθεί το δουβλίνο τρία που μετατρέπει την ελλάδα σε αποθήκη ψυχών καθιέρωση της ρήτρας κατανομής προσφύγων σε όλα τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης ανάλογα με το αεπ την έκταση και τον πληθυσμό κάθε κράτους μέλους. πέμπτον να ενισχυθεί οικονομικά η ελλάδα για καλύτερη φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων. τέλος πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι η διαφύλαξη των ελληνικών συνόρων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της ελλάδας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα προστασίας των ελληνικών συνόρων δεν πρόκειται να τα εκχωρήσουμε στην τουρκία ή στην ευρωπαϊκή ένωση. ευχαριστώ. Παρακαλώ και λυπούμε αν σας πρόφερα το όνομα λάθος. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Πρόεδρε, κύριε Τούσκ. Προσπίζεστε την ε, ε, καλή φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους διαδρόμους των Ηνωμένων Εθνών. Και όμως στο δρόμο για την Ευρώπη χάνουν τη ζωή τους ακόμη και παιδιά. Εσάς τώρα σας νοιάζει να σώσετε τη φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναρκισισμός είναι αυτό. Όταν διαπράττουμε το ένα λάθος μετά το άλλο. Όχι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο που δεν μπόρεσε να προτείνει ένα ε, γενικό σχέδιο που να αντιμετωπίζει όλες τις πτυχές προβλήματος. Αποτύχατε κύριε Τούσκο. Και επίσης πάντοτε Μιλούμε για τις αξίες όταν θέλουμε να προδώσουμε κάτι. Κύριε Τούσκ, τα εξωτερικά σύνορα σας ενδιαφέρουν. Ούτε οι αξίες, ούτε η αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δυστυχώς ούτε και η αποτελεσματικότητα. Αυτή είναι η κατάσταση. Ευχαριστώ κύριος Χρυσόγονος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συζητούμε για πολλωστή φορά στην αίθουσα αυτή για το προσφυγικό πρόβλημα ως εάν η προσφυγοποίηση των ανθρώπων να ήταν ένα φυσικό φαινόμενο όπως η ηλιοφάνεια ή η βροχή δεν είναι φυσικό φαινόμενο είναι αποτέλεσμα των πολέμων και για τους πολέμους αυτούς ιδίως για τον πόλεμο στη συρία που διαρκεί ήδη τέσσερα και πλέον χρόνια συνυπετιότητα έχουν και οι κυβερνήσεις δυτικών κρατών τόσο των ηνωμένων πολιτειών όσο και ορισμένων μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών που δεν μπορούν να απαλλαγούν από την έμονη ιδέα ότι πρέπει να επιβάλλουν σε όλο τον κόσμο ακόμα και εκτός της δύσης καθεστώτα της αρεσκίας τους είναι φανερό ότι η προσπάθεια της δύσης να ενισχύσει την συριακή αντιπολίτευση για να ανατρέψει το καθεστώς ασαντ έχει αποτύχει και έχει οδηγήσει στην ενίσχυση και στο θέργεμα του φαινομένου του ισλαμικού κράτους. πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν υπάρχει λύση στη συρία χωρίς τον ασαντ και να προχωρήσουμε ρεαλιστικά για να ξεριζώσουμε το ισλαμικό κράτος για να σταματήσει η προσφυγοποίηση. Η κυρία Λούνα της ένα λεπτό. Έλα, Ουλρίκε. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής του Συμβουλίου. 22 Συμβουλίου ήταν καλό το, το Συμβούλιο των Εσωτερικών ε, και της Δικαιοσύνης αποφάσισε την ε, κατανόμη όλων των προσφύγων σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεσμικά μάλιστα είναι καλό μήνυμα, μήνυμα αλληλεγγύη η απόφαση αυτή. Αλλά πρέπει και να υλοποιηθεί τώρα. Χρειάζεται συμμαχία του ανθρωπισμού, της ανθρωπιάς που να λειτουργήσει, να δράσει υπέρ των ανθρώπων, των γυναικών και των ανδρών που προσπαθούν να ξεφύγουν από τις βόμβες του Ασάτ και από τους ε, μαχητές του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους. Πρέπει να πούμε ναι θα τα καταφέρουμε και γι' αυτό είναι απαραίτητο να καταργηθεί το Δουβλίνο. Πρέπει να βρεθούν νόμιμοι τρόποι μετανάστευσης, να μπαίνουν οι άνθρωποι αυτοί σε κάποιους πραγματικούς καταβλισμούς υποδοχής και όχι στα πλοία της Frontex. Ε, όταν έρχεται ο Ερντογάν λοιπόν για να συνομιλήσει και λησμονούμε προκειμένου να συστήσουμε το θέμα των προσφύγων, την, τον αυταρχισμό του και την καταστολή και το πάρκο Γκεζί και τους Κούρδους και όλα τα άλλα προβλήματα, κύριε ε, τους χρειάζεται μια ε, θαραλέα πολιτική. Ας μην υποκύπτουμε στους λαϊκιστές. Όπως και να λέγονται, Φίντες λέγονται, φόνασιονά λέγονται, όπως και να λέγονται, δεν πρέπει να υποκύψουμε στους λαϊκιστές. Βίμπεργκερ ένα λεπτό. Πρόεδρε. Αισθάνομαι κατάπληξη. Έχω την εντύπωση ότι βρισκόμαστε μέσα σε μια σφαίρα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σαν να μην έχουμε σχέση με την πραγματικότητα. Μιλάτε για αλληλεγγύη. Μα για μένα η αλληλεγγύη έπρεπε να έχει εκφραστεί έναντι του παγκόσμιου επισητιστικού προγράμματος, επί παραδείγματι, όταν μιλούσαμε για βοήθεια για τους ανθρώπους που λιμοκτονούν. Η αλληλεγγύη είναι τα χρήματα που πρέπει να δοθούν σε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη. Ενώ τώρα την αλληλεγγύη και τα χρήματα τα δίνουμε στους μετανάστες. Στη Σουηδία, τη χώρα μου, μιλούμε για ενσωμάτωση όλων αυτών που έρχονται. Πρέπει να τους ενσωματώσουμε, λέμε. Χρόνια τώρα το λέμε στη Σουηδία. Δεν λειτουργήσε όμως αυτό. Έχουμε 55 ζώνες στις οποίες δεν ισχύει το δίκαιο και το κράτος στην ε, Σουηδία. Δεν έχουμε αρκετή στέγη να προσφέρουμε. Και μάλιστα έχει φτάσει η Σουηδία να διαρωτάται αν πρέπει να φτιάξει έναν πρώτο καταβλισμό προσφύγων σε αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ Μπάλτσου. Τελευταία παρέμβαση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος Γιούνκερ πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δείχνει έκπληκτος που οι πρωθυπουργοί δεν έλαβαν ομόφωνη απόφαση για τις ποσοστώσεις. Για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους. Ναι, αυτή είναι η απάντηση. Κάποιες ε, χώρες και κυβερνήσεις λαμβάνουν υπόψη το τι θέλουν οι πολίτες τους. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών επέκρινε την Ουγγρική κυβέρνηση χωρίς να έχει κανένα τέτοιο δικαίωμα για την πράσπιση των σύνορων μα. Όμως, περισσότερες ε, κυβερνήσεις συμφωνούν με την έγκριση αυτού του φράχτη, αυτού του τείχους. Ο κύριος Τούσκ μας ζήτησε περισσότερη ελληνική και περισσότερη Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι η πιο ανοιχτή κοινωνία, η πιο ανεκτική και πιο ανοιχτόμυαλη. Όμως υπάρχουν προκλήσεις και πιέσεις κατά της δημοκρατίας. Εάν είναι κανείς δημοκράτης θα πρέπει να σέβεται και το τι θέλει ο πληθυσμό τη Ευρώπη και με δημοψηφίσματα. Ευχαριστούμε. Τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γιούνκερ, έξω ονόματο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όντω, η Ευρώπη δεν μπορεί να υποδεχθεί όλου του δυστυχεί του κόσμου στην επικρατεία τη. Όμω, πρέπει να ασχοληθεί με τη δυστυχία του κόσμου η Ευρώπη ολόκληρη. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε ουδέτεροι ούτε αμετακίνητοι χωρίς να αντιδρούμε όταν βλέπουμε τόσες αδικίες, όταν τόσα σοβαρά γεγονότα συμβαίνουν αλλού στον πλανήτη μας. Όντως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα γενεσιουργά αίτια, τις πηγές του προβλήματος της μετανάστευσης. Κάποιοι το κάνουν ήδη να αποτέσω φορό τιμή στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν περιέκοψαν την και του βοήθεια. Είναι πολλοί, είναι περισσότεροι. Και επίση να αποτέσω φορό τιμή σε όσου σκοπό έχουν να αυξήσουν τη βοήθεια που προσφέρουν ε, στην κατεύθυνση τη ανάπτυξη. Και θα επικρίνω τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που μείωσαν τη συνεισφορά του στον ίδιο σκοπό την ανθρωπιστική βοήθεια. όσους μείωσαν τη συνεισφορά τους στο Παγκόσμιο Επισκεπτικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών. Ε, τα κράτη-μέλη επίσης που μείωσαν τη συνεισφορά τους για τη λειτουργία της επαθυσαρμοστίας για τους πρόσφυγες. Αν θέλουμε λοιπόν να μιλούμε για τα αίτια, θα πρέπει να μιλούμε και για όσους συνεισέφεραν στο να ε, διωγκωθεί αυτή η σωρία προβλημάτων που οδηγούν τους πρόσφυγες να έρχονται στην Ευρώπη. Και για να τα λέμε και όλα ξεκάθαρα εδώ, θα πρέπει να είμαστε περήφανοι. Διότι όσοι είναι δυστυχείς έρχονται προς την Ευρώπη. Η Ευρώπη στα μάτια τους φαίνεται ως ένας τόπος όπου ο ήλιος λάμπει περισσότερο από ό,τι γιατί δεν πάνε στην Κίνα. Γιατί δεν πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί δεν πάνε στις χώρες του κόλπου. Θα πρέπει τώρα να ζητάμε και συγνώμη που όλος ο πλανήτης μας βλέπει ως τον τόπο όπου ο καιρός είναι καλύτερος και είναι πιο ωραία να ζει κανείς. Θα πρέπει να είμαστε περήφανοι, αλλά θα πρέπει να μπορέσουμε να διαχειριστούμε και, την, και τον τεράστιο αυτό όγκο, το τεράστιο κύμα προσφύγων και το κάνουμε ήδη η σωστή απάντηση για την μετανάστευση δεν είναι η οικοδόμηση τυχών. Οι πρόσφυγες, οποιοδήποτε, οι οποιοδήποτε δυστυχείς, θα βρίσκουν έναν τρόπο να φτάνουν στην επικράτεια της Ευρώπης. Ό,τι και να κάνουμε. Είτε χτίσουμε τύχη, ε, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν θα λύσουμε το πρόβλημα. Όσοι χτίζουν τύχη τουλάχιστον θα πρέπει να προσέχουν τι λένε ταυτόχρονα ε, με το αρχιτεκτονικό τους έργο. Μην ξεχνάμε ότι τα λόγια τους μιλάνε σε όσους τους ακούν. Πώς μπορούμε να λέμε ότι οι πρόσφυγες είναι οικονομικοί πρόσφυγες χωρίς να υψώνονται φωνές διαμαρτυρίες. Πού το ξέρετε υπάρχουν κάποιοι που διαφεύγουν από τη χώρα τους γιατί διώκονται. Να μην μπερδεύουμε λοιπόν ε, διαφορετικά πράγματα. Ναι, υπάρχουν οικονομικοί πρόσφυγες. Εάν ζούσατε στις δικές τους συνθήκες διαβίωσης, τι θα κάνατε στη θέση τους. Δεν έχουν το ίδιο δικαίωμα να παραμένουν στην Ευρώπη. Εντάξει, όμως ας μην αναφερόμαστε σε αυτούς τους δυστυχής σαν να επρόκειτο για εγκληματίες και οργανωμένες συμμορίες. Είναι όλοι δυστυχεί. Είπα ότι η οικοδόμηση τυχών δεν είναι η καλύτερη απάντηση και θα προσθέσω το εξής. Γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να γύρουν τύχη μεταξύ των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ χωρών. Γιατί μεταξύ ε, κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση η οικοδόμηση τυχών δεν μπορεί πλέον να συμβαίνει. Γιατί δεν ενοχλεί πια. Πώς μπορεί εν έτη 2015 κάποιοι να χτίζουν τύχη μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. Πρέπει σε αυτή την περίπτωση ανοιχτά να επικρίνουμε τις κυβερνήσεις που τολμούν να κάνουν τέτοια αρχιτεκτονικά έργα. Κάποιοι από σας επικρίνατε με δρυμύτητα την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν λαμβάνει τις σωστέ αποφάσει. Να θυμίσω εδώ ότι οι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στι 23 Σεπτεμβρίου μόλις ελήφθησαν και τα κονδύλια ε, που θα ακολουθήσουν τις αποφάσεις αυτές του Συμβουλίου θα ψηφιστούν από το Κοινοβούλιο στι 15 Οκτωβρίου. Νομίζω ότι αυτή τη φορά δράσαμε ταχύτητα. Συμβούλιο, Επιτροπή και Κοινοβούλιο μαζί και μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Αν ήμασταν πάντοτε τόσο ταχεί και τόσο άμεση, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή θα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Επικρίνεται τα κράτη-μέλη. Εντάξει, αλλά λέτε πάντοτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν είναι σωστό. Μη λέτε συνέχεια η Ευρώπη και η Ευρώπη και η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μην τους βάζετε όλους στο ίδιο καλάθι. Ε, να λέτε κάποια κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση να λάβουν τις αποφάσεις που θα έπρεπε. Μην επικρίνετε την Ευρώπη, επικρίνετε τα κράτη-μέλη. Αυτά που μας εμποδίζουν να δράσουμε. Και σε κάθε περίπτωση μην κριτικάρετε το φίλο μου τον κύριο Τούσκ. Είμαι μάρτυρας του πώς εκτελήχθηκαν οι σύνοδοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εάν κάποια κάτι μέλη εμποδίζουν τον πρόεδρο του Συμβουλίου να προχωρήσει με την ε, ταχύτητα που θα ήθελε να έχει το ε, Συμβούλιο. Μην επικρίνετε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που κάνει ό,τι μπορεί για να προχωρήσουν τα πράγματα. Ε, να επικρίνετε αυτά τα κράτη-μέλη. Αυτούς που δυσκολεύουν την κατάσταση. Επιπλέον, θα πρέπει πάντως, πάντοτε να επανερχόμαστε σε ένα θέμα που είναι μείζονο σημασία. Εμένα ε, μου κινεί την περιέργεια το γεγονό ότι ο θρησκευτικό παράγοντα και ο φιλοσοφικό παράγοντα ε, λαμβάνουν στην Ευρώπη διαστάσει που δεν του αρμόζουν. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε μια επικράτεια αυστηρό χριστιανική. Δεν μπορούμε να λέμε ότι στην επικράτειά μα δεν θέλουμε να έχουμε άλλα θρησκευτικά δόγματα. Δεν είναι έτσι η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι η ήπειρος της ανεκτικότητας. Δεν πρέπει να υπάρχει ανοχή ως προς την ε, έλλειψη ανοχής. Αυτό πρέπει να το λέμε διαρκώς. Και κατά τα άλλα... Θέλω να πω και το εξής ως απάντηση. Μην παρετήσετε από το δικαίωμα να πείτε κύριε Τούσκο, εχτε... δεν μπορείτε να λέτε ότι κάναμε μια συζήτηση γύρω από ένα φλιτζάνι καφέ. Όχι, συζητήσαμε σοβαρά θέματα που αφορούν τους πρόσφυγες. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Αλλά και άλλα ζητήματα συζητήσαμε βέβαια. Φυσικά και είναι φυσικό να δώσουμε το χέρι στον κύριο Ερντοάν, αλλά φυσικά και συζητήσαμε άλλα προβλήματα. Το είπε και ο πρόεδρος, πράγματα που μας διαφοροποιούν. Αλλά η Τουρκία είναι ασφαλές κράτος, ανήκει σε αυτόν τον κατάλογο. Αυτοί που λένε ότι θα πρέπει να συμβαίνει το αντίθετο, πρέπει και να δεχθούν τις συνέπειες αυτής της επιλογής. Γιατί αν δεν ανήκει στα ασφαλή κράτη η Τουρκία, τότε πρέπει να, να διακοπούν αμέσως, να καταθέσουν το αίτημα για διακοπή των συνομιλιών για ένταξη. Στο βαθμό όμως που χρειαζόμαστε και τη βοήθεια της Τουρκίας και στο βαθμό που υπάρχει αρμονική συνεργασία της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο βαθμό που θεωρούμε ότι δεν πρέπει να διακοπούν οι συνομιλίες παραμένει η Τουρκία και στο βαθμό αυτόν παραμένει η Τουρκία στον κατάλογο των ασφαλών των ασφαλών κρατών. Αλλά μην νομίζετε ότι ανταλλάξαμε μόνο αυρότητε με τον κύριο Ερτογάν. Αλλά δεν μπορούμε και να σμονούμε ότι έχει υποδεχθεί 2,2 εκατομμύρια πρόσφυγε στην επικράτειά τη. Είναι δυνατόν να ισχυριστεί κανεί ότι δεν είναι τεράστια αυτή η επιβάρυνση και ο κόπο. 2,2 εκατομμύρια. Για σκεφτείτε ποιο θα δεχόταν με αλληλεγγύη στην Ευρώπη 2,2 εδώ δυσκολευόμαστε για τι 160.000. Η Τουρκία έχει 2,2 εκατομμύρια υποδεχθεί στην Τουρκία. Για να μην μιλήσω για τον Λίβανο και την Ιορδανία. Που έχουν πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση αναλογικά του πληθυσμού τους. Ας είμαστε λοιπόν ειλικρινείς. Είμαστε στην αρχή μιας μακράς διαδικασίας. Χρειαζόμαστε όμως ακριβώς γι' αυτό λόγο ένα μόνιμο σύστημα αναδιανομής στην Ευρώπη. Γι' αυτό χρειάζεται και ένα νόμιμο σύστημα της μετανάστευσης στην Ευρώπη. Εγώ προέρχομαι από μικρή χώρα, το Λουξεμβούργο για δεν το γνωρίζει. Εγώ μεγαλώνοντας έκανα παρέα με Ιταλούς, με Πορτογάλους, και το Λουξεμβούργο είναι από τα πιο πλούσια κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρί του Πορτογάλου και του Ιταλού, το μικρό αυτό κρατήδιο δεν θα είχε γίνει αυτό που έγινε εν τέλει. Γιατί η μετανάστευση φέρνει πλούτο. Σα ευχαριστούμε Πρόεδρε Γιόνκερ και τώρα ο Πρόεδρος Τούσκ και θα σα διαδεχτεί, θα με διαδεχτεί ο κύριος Ταγιάννης στην ε, Προεδρία. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Ζαν Κλοντ για την υποστήριξή του. Βεβαίω όμω το αναμένω ότι θα δεχθώ κριτική όταν έρχομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν έρχομαι να λάβω το χειροκροτήματα. Τα δουλειά μου είναι να ακούω την κριτική σα. Και βεβαίω η κριτική αυτή πρέπει να είναι αυστηρή. Ε, για να είμαστε σωστοί στην άσκηση της πολιτικής όπου όλα αυτά τα θέματα πρέπει να συζητούνται ανοιχτά. Καλωσορίζω τη συζήτηση γιατί πιστεύω ότι μετά από τη συζήτηση αυτή όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι το πρόβλημα αυτό, αυτό το θέμα συνεχίζει να διχάζει τους Ευρωπαίους και καταλαβαίνω γιατί. Στο εσωτερικό των κρατών μελών επίσης είναι διχασμένη η κοινή γνώμη. Όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω όμως ότι σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να ακολουθήσουμε μια πιο κοινή πολιτική. Πολύ περισσότερο από ότι ε, θα μπορούσε κανείς να το πει πριν από λίγες εβδομάδες. Δεν έχω ψευδεστήσεις. Και χωρίς αμφιβολία, τίποτα δεν θα είναι εύκολο όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Πρώτα απ' όλα εξαιτίας του μεγέθους του προβλήματος. Που είναι μεγαλύτερο από ποτέ. Και γι' αυτό το λόγο δημιουργεί τέτοιες παθιασμένες συγκρούσεις. Και όχι μόνο στο Ευρωκοινοβούλιο όπως είπα. Πρώτα απ' όλα, Θέλω να τονίσω το εξή. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια μοναδική κατάσταση εξαιτία του μεγέθους τη. Σήμερα μιλούμε για περίπου 70 εκατομμύρια εκτοπισμένους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε περιοχές οι οποίες βρίσκονται περιμετρικά της Ευρωπαϊκής Υπήρου. 70 εκατομμύρια. Στην Αφρική, στην Ασία. Τρία εκατομμύρια Αφγανοί έχουν εγκαταλείψει τις αιστείες τους και πηγαίνουν προς άλλες χώρες, στο Πακιστάν, στο Ιράν, στο Ιράκ, στην Τουρκία. Κάποιοι από αυτούς έχουν ήδη φτάσει στην Ευρώπη. Τρία εκατομμύρια Αφγανοί λοιπόν πρέπει να ξέρουμε, πρέπει να αντιληφθούμε ότι αν όχι για όλους, αλλά πάντως για τη μεγάλη πλειονότητα αυτών των τριών εκατομμύριων Αυγανών, η τελικός προορισμός θα ήταν η Ευρώπη, ο επιθυμητός. Οι εσωτερικά εκτοπισμένοι στη Συρία είναι τρία εκατομμύρια επίσης. Τρία εκατομμύρια Σύριοι στην Ιορδανία, στην Τουρκία. Εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες από την Ιεμένη. Για όλους αυτούς τους λόγους η λύση δεν είναι εύκολη. Για όλους αυτούς τους λόγους ανησυχούμε πολλοί από εμάς στην Ευρώπη. Και επίσης για αυτούς τους λόγους υπάρχει και ο φόβος στην Ευρώπη. Είναι λογικό κατά μία έννοια. Μπορούμε να το περιμένει κανείς. Δεν είναι καινούριο πρόβλημα το προσφυγικό. Αυτό που είναι καινούριο είναι το, η κλίμακα του προβλήματος. Αυτή η μαζική έξοδος είναι ε, το καινοφανές. Υπάρχουν κάτι που δεν έχουν ε, την εμπειρία ε, στο παρελθόν να έχουν αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό έχει γίνει τόσο έντονη η δημόσια συζήτηση. Δεν μπορώ να δεχθώ την θέση που λέει ότι η πλειονότητα των προσφύγων είναι στην πραγματικότητα μετανάστες. Πρώτα απ' όλα, στη σημερινή πραγματικότητα είναι σχεδόν αδύνατον να κάνει κανείς τη διάκριση μεταξύ προσφύγων και μεταναστών. Γιατί όλοι τους εγκαταλείπουν τις αιστείες τους εξαιτίας πολέμου, πείνας, ανέχειας ταυτόχρονα για αυτούς τους λόγους και τους τρεις αυτούς λόγους ταυτόχρονα και από τη Συρία και από το Αφγανιστάν και από παντού. Αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος που περιπλέκει τα πράγματα. Γιατί όλους πρέπει να τους θεωρήσουμε, σχεδόν όλους, πρέπει να τους θεωρήσουμε πιθανούς τον Δεύτερον, ένας ακόμα λόγος που δεν μπορούν να βρεθούν εύκολες λύσεις το, η άνοπλη σύγκρουση στην Σύρια. Μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμια σύγκρουση, γιατί έχουν εμπλακεί δυνάμεις μεγάλες του πλανήτη. Η κατάσταση είναι ήδη πολύ επιδεινωμένη και μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο προσφύγο κύμα από την Συρία. Όπως είπα, οι εκτιμήσεις μιλούν για 3 εκατομμύρια επιπλέον νέους πρόσφυγες. Να έχουν φύγει από το Χαλέπι και τις γειτονικέ περιοχές. Τρίτον, ένας ακόμας λόγος που η κατάσταση είναι δύσκολη. Οι χώρες με τις οποίες πρέπει να συνεργαστούμε δεν είναι εταίροι με τους οποίους εύκολα μπορεί να συνεργαστεί κανείς. Πρέπει να συνεργαστούμε για παράδειγμα με την Τουρκία. Καταλαβαίνω το σκεπτικισμό, καταλαβαίνω τις ανησυχίες των συναδέλφων που ε, αναφέρονται στην Τουρκία. Αλλά εάν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα είναι απολύτως απαραίτητο να συνεργαστούμε με την Τουρκία. Είναι κρίσιμος εταίρο. Μπορούμε να τους κάνουμε μαθήματα. Αυτό θέλουμε. Ή να τους πάρουμε μαζί μας, τους Τούρκους, και να συνεργαστούν μαζί μας για την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Και κατανοώ τη δραματικότητα του διλήμματος που σας θέτω. Αλλά αυτό είναι το δίλημα σήμερα. Το δίλημα που πρέπει να απαντήσουν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης είναι πώς θα συνεργαστούμε με την Τουρκία μιας και δεν γίνεται αλλιώς. Και υπάρχουν και άλλοι εταίροι ακόμα πιο δύσκολοι από την Τουρκία. Θα έλεγα ότι όσον αφορά τις γειτονικέ χώρες της Ευρώπης η Τουρκία είναι από τους πλέον εύκολους εταίρους Γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι και στην επόμενη ε, σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα συζητήσουμε εις βάθος το προσφυγικό. Και ελπίζω ότι η συζήτηση που έγινε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εμπλεύσει τις ε, ορισμένους ηγέτες, ορισμένα κράτη-μέλη να αλλάξουν τη θέση τους και νομίζω όλοι καταλάβατε τι εννοώ. Και μια ερώτηση από Πολωνό βουλευτή, τον κύριο Όλμπρεχτ. Τι μπορούμε να κάνουμε ή τι πρέπει να κάνουμε. Χώρια και μαζί, ως πρώτη μέλη. Ένα πράγμα είναι σαφές σήμερα. Κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί μόνο του να υποδεχθεί όλους τους πρόσφυγες που έρχονται. Γι' αυτό χρειάζεται σύστημα αναδιανομής. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι στα εξωτερικά μας είναι ώρα κανείς πάλι δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις ροές που φτάνουν. Αυτά είναι λοιπόν ζητήματα τα οποία απαιτούν κοινή αντιμετώπιση και προσέγγιση. Ας σταματήσουμε λοιπόν να καταγγέλουμε και να κατηγορούμε ένας τον άλλον. Γι' αυτό πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη προστασία των εξωτερικών συνόρων. Είναι σαφές πια σήμερα νομίζω ότι το άνευ προηγουμένου αυτό βάρος και ευθύνη ξεπερνάει τις δυνατότητες ή ουδήποτε κράτους μέλους. Μπορεί αυτό να πρέπει να σημαίνει ρήξη, επανάσταση διανοητική για μας, να, να αλλάξουμε τρόπο σκέψης. Αλλά πρέπει να το πράξουμε. Πρέπει να αναλάβει το μέρος της ευθύνης, της προστασίας των εξωτερικών συνόρων η Ευρώπη. Όπως και για τα θέματα της αναδιανομής, τα λεγόμενα hot spots, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα αντιμετωπίσει η Ευρώπη ενωμένη και να βοηθήσει και τις χώρες εκτός των σύνορων της για τον προσδορισμό λύσεων. Αυτό θα είναι απαραίτητο και χρήσιμο για όλα τα θεσμικά όργανα. Σας ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ και εγώ, Πρόεδρε Τούσκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Γιούνκερ, για τις τοποθετήσεις σας εδώ, αλλά πάνω απ' όλα για την στράτευσή σας. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση.